Okay, good morning, dear colleagues, ladies... Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε. Είναι η δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας αυτή τη βδομάδα. Και είμαστε στα σημεία 7 και 8. Πρόκειται για μια κοινή συζήτηση που θα κάνουμε όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη της Γενέβης της Συμφωνίας της Λισαβόνας. Έχουμε δύο εισηγητές. Ο ένας για την προσχώρηση και ο άλλος για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θα δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στον κύριο Χάνσεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως βλέπετε από την παρουσία, πολύ ενδιαφέρονται για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Όμως, είναι ένα σημαντικό θέμα για να μιλήσουμε πιο σοβαρά, αποτελεί μέρο της ε, Συμφωνίας της Λισαβόνα του 1958, που είναι μια διεθνής καταχώρηση για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Οι διεθνείς οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος. Σήμερα όμως μπορούμε. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα διότι η συμφωνία αυτή ενισχύει την προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε τα μέσα κύρωσης που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει και θέτουν το ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της εφόσον έχει ολοκληρωθεί προσχώρηση. Η ομάδα μου λοιπόν καλωσορίζει το θέμα αυτό γιατί πάντα το ΕΛΚ ήταν υπέρ το, της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κερδίζουν το ψωμί τους και να αναπτυχθεί ύπεθρος. Πρόκειται επίσης για την προστασία της ευρωπαϊκής ποικιλομορφία μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μόνο 7 χώρες μέλη συμμετέχουν στη Συμφωνία της Λισαβόνας τώρα ως κράτη. Η προσχώρηση αυτή όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη της Γενέβης θα βοηθήσει την προστασία των γεωγραφικών αδείξεων σε διεθνές πλαίσιο. Πολλά είναι τα ωφέλη για το εμπόριο, διότι η πράξη της Γενέβης προστατεύει περισσότερο από τη Συμφωνία TRIPS στα πλαίσια του ΠΟΕ. Οπότε η ενίσχυση αυτή μέσω της πράξης της Γενέβης είναι πολύ σημαντική αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων, διμερός, μπορεί να είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ, κοστίζει πολύ και δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλύτερη η πράξη της Γενέβης Εφόσον αναγνωρίζονται οι γεωγραφικές ενδείξεις μέσω της πράξης της Γενέβης, πιστεύω ότι πετυχαίνουμε πολύ καλύτερη προστασία. Θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που κοινοποιούμε στο, στην πολυμερή καταχώρηση. Και μετά από όλα αυτά τα επιχειρήματα, ο συντάκτης γνωμοδότησης για την προσχώρηση της Ένωσης φυσικά και συστήνω την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι πολύ καλά ισορροπημένη. Έχω δύο τροπολογίες που έχω υποβάλει, οι οποίες επαναλαμβάνουν ότι το κείμενο θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως στη Συμφωνία TRIPS για οτιδήποτε καινούριο προκύψει στον ΠΟΕ και δεύτερον λέω ότι η πράξη της Γενέβης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διμερώς να προστατεύει τις γεωγραφικές της ενδείξεις σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών βάσει των συνθηκών της αγοράς όπως προκύπτουν κάθε φορά. Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι η πολιτική μας γεωγραφικών ενδείξεων έχει αποτελέσει αντικείμενο ε, επιθέσεων τελευταία με κάποιες εξαιρέσεις από τα τυριά για παράδειγμα στην αγορά των ΗΠΑ και του Μεξικού παρόλο που δεν έχει να κάνει απευθείας με τις γεωγραφικές ενδείξεις των ε, τυριών παρόλα αυτά καλό θα ήταν να ενισχύσουμε την προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων για να προστατεύσουμε μικρής κλίμακας παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και ό,τι σχόλια έχετε να κάνετε είναι ευπρόσδεκτα. Πρόεδρος, ωραία. Δεύτερη έκθεση, Τιτσιάνα Μπεγκίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε ο Απλώς θα περιλάμβανα ίσως κάποια επιπλέον στοιχεία σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, προϊόντων που δεν είναι γεωργικά ή προς διατροφή και προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις αλλά θα φροντίσουμε να υποβάλουμε σχετική τροπολογία. Σε ό,τι αφορά το να συμφωνήσουμε ή όχι, εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσέξουμε την εξή ανάγκη. Είναι χιλιάδε οι γεωγραφικέ ενδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι όλα προϊόντα τα οποία προέρχονται από ε, αιώνε παράδοση, όπω το προσώτο τη Πάρμα ή η Παρμεζάνα, η Παρμεζάνο Ρετζάνο. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει ε, πολύ έγευστα προϊόντα πολύ χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να προστατεύσουν τον τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα η χώρα μου είναι αυτή που ε, ωφελείται περισσότερο από αυτή την προστασία και είναι και μοντέλο με πάνω από 1.800 ε, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και αξία ε, πολλών δις ευρώ. Είναι λοιπόν σημαντικό να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα προϊόντα αυτά. Από το 2015 η Συμφωνία της Λισαβόνας έχει καλύψει και τις γεωγραφικές ενδείξεις υπό ευρία έννοια. Και αυτό που υποβάλλεται σήμερα στο Κοινοβούλιο είναι σημαντικό, διότι η Ένωση θα συμβληθεί στην συμφωνία αυτή. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφή. Χάρη σε αυτό το εργαλείο θα έχουμε καλύτερη προστασία τη γεωγραφική μα ενδείξη με μία μόνο καταγραφή. Μία μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη αλλά και στι υπόλοιπε ε, χώρε που έχουν συνυπογράψει. Αυτή τη στιγμή 7 ευρωπαϊκέ χώρε είναι μέρο τη ε, ε, σύμβαση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν οι γεωγραφικέ ενδείξει να προστατευτούν και να, γίνει, να συμπληθούν οι υπόλοιπε χώρε σε παράρτημα θα πρέπει να δούμε το σύστημα προστασίας που προσφέρεται από αυτό το εργαλείο χωρίς να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε διαφορετικές ε, γεωγραφικές ενδείξεις και λιγότερα αποτελεσματικές. Η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα της Λισαβόνας είναι πολύ ε, σημαντική για τις γεωγραφικές ενδείξεις γενικώ και γι' αυτό εύχομαι γρήγορα να εγκριθεί από αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης κύριος Grazie Presidente. Come ricordato da entrambi i relatori, il Parlamento... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εδώ πρέπει να αποφανθούμε για, την, ε, για το κατά πόσο να συμβληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη τη Γενέβη και τη Συμφωνία τη Λισαβόνα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, όπου ο ΠΟΕ για την προστασία των, των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία και νομική προστασία θα αποφασίσει για την εφαρμογή όχι. Είναι επιπλέον βήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση τη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στι τρίτε χώρε με μεγαλύτερη διάδοση της φιλοσοφίας που συνοδεύει το εργαλείο αυτό. Δηλαδή το να αξιοποιηθεί η χαρακτηριστική ποικιλομορφία των τοπικών προϊόντων, περιφερειακών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των παραδοσιακών ε, βιοτεχνικών παραγωγών και των προϊόντων που προκύπτουν, καθώς και την ενίσχυση του δεσμού παραγωγού και καταναλωτή, που λαμβάνει αξιόπιστες πληροφορίες για τον τόπο και τη μέθοδο παραγωγής. Εφόσον προσχωρήσουμε στη συμφωνία αυτή, θα ε, ενισχυθεί το σύστημα που ε, στο πλαίσιο των εμπορικών τη συμφωνιών διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα οποία προσπαθούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητα στην αγορά τρίτων χωρών. Και θα συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση τη παραποίηση και τη ε, παράνομη χρήση ε, καταγεγραμμένων γεωγραφικών ενδείξεων, των οποίων είναι θύματα κάποια αγροτικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για εξαγωγέ πολύ σημαντικέ για την ευρωπαϊκή οικονομία που αξίζουν πάνω από 11 και είναι το 15% των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον τομέα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και των ποτών. Ε, σε σχέση με την πράξη της Γενέβης, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Χάνσεν για το σχέδιο γνωμοδότησής του και να εκφράσω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Πρώτον, πιστεύω ότι ο κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποβάλει στον Διεθνή Οργανισμό θα πρέπει αυτομάτω να περιλαμβάνει τι γεωγραφικέ ενδείξει που ήδη έχουν καταγραφεί από 7 κράτη-μέλη στου αρμόδιου φορεί προτού συμπληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μέτρο είναι απαραίτητο για να υπάρξει συνέχεια στην προστασία. Έπειτα θεωρώ ότι δεδομένη της ε, ενδεχόμενης καταγραφή ε, των ε, προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να προβλέψει έναν μηχανισμό περιοδικής και συστηματικής αξιολόγησης με τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει ένα συνεχής διάλογος με τους αρμόδιους φορείς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ των προστατευόμενων γεωργικών προϊόντων και αυτών που δεν είναι γεωργικά. Υπάρχουν προϊόντα που σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό προστατεύονται ω προ τι γεωγραφικέ του ενδείξει, 14 προ 20, ενώ υπάρχουν άλλα κρατημέλη όπου ε, η προστασία γίνεται μόνο από του αρμόδιου φορεί τη Γενέβη. Αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, θα έπρεπε να έχει εξεταστεί ήδη και να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος αυτό από τον περασμένο Γενάρη. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε καλή συνεργασία για την έγκριση και των δύο προτάσεων. Εν... Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Σχάκιο. Sorry, I wasn't paying attention. Συγγνώμη, δεν πρόσεχα. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους της ομάδας μου για τις γεωγραφικές ενδείξεις Ευχαριστώ. Um, Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις. Ούτε έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κλάους Μπλάνκ από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ε, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την θετική στάση απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν. Για πάνω από 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί επιτυχημένη πολιτική προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων τόσο στην εσωτερική της αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. Αυτή η πολιτική παρέχει σαφή πλεονεκτήματα στους επιχειρούντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχοντας κάνει λοιπόν μεγάλες προσπάθειες και έχοντας επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στην Συμφωνία της ε, Λισαβόνας, η οποία κατέληξε και στην έγκριση της πράξης της Γενέβης στο συνέδριο του 2015 του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας προτείνουμε πλέον να προσχωρήσουμε στην πράξη αυτή. Είναι σημαντικό να καταστεί μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθώς και για την αξιοποίηση του Παγκόσμιου Θεματολογίου για την Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Αυτή είναι και η μόνη εύλογη προσέγγιση. Η πολιτική αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με, τους, με τα συμφέροντα των εμπλεκομένων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τους πλήττει ούτε τους επιβαρύνει οικονομικά ή διοικητικά. Επίσης, συνάδει και με τις πολιτικές και τη στάση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποκλειστεί θεωρώντας μάλλον της ε, αποκλειστικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Η νέα πράξη της Γενέβης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην παγκόσμια στρατηγική μας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων παγκοσμίω. Επιπροσθέτως προς τις ε, ε, διμερείς βεβαίως εμπορικές συμφωνίες με απότερο σκόπο την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Το να καταστεί λοιπόν η Λισαβόνα ανοιχτή σε διεθνείς οργανισμούς ήταν μία, ένας από τους στόχους της διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διπλωματική συνδιάσκεψη, θα συμβάλλει στην προστασία των ενωσιακών γεωγραφικών ενδείξεων μέσω της κατάρτισης ενός πολυμερούς μητρώου γεωγραφικών ενδείξεων και θα συμβάλλει ιδίως στην ε, προστασία ίνων και ινοπνευματοδών αλλά και άλλων γεωργικών ε, προϊόντων. Θα συμβάλλει στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε πολυμερές και διμερές επίπεδο με ε, εξειδίκευση σε διάφορες χώρες. Πολλά μέλη του WIPO ενδιαφέρονται για την κατάρτιση ενός ευρύτερου μηχανισμού προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων και αυτό αποδεικνύεται και με την προσχώρηση και άλλων χωρών στην πράξη της Γενέβης όπως της Ρωσίας και της Κίνας. Θα υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει. Οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποκτήσουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω αυτής της πράξης της Γενέβης. Και αυτό είναι ε, ε, ιδιαίτερα σημαντικό αν προσχωρήσουν και άλλες χώρες στην πράξη της Γενέβης, όπως είναι οι χώρες ΑΖΕΑΝ, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Τουρκία, καθώς και διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι οι δύο οργανώσεις της Αφρικής για την διανοητική ιδιοκτησία. Η δημιουργία ενός πολυμερούς μητρώου γεωγραφικών ενδείξεων θα βοηθήσει στην προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και στην επίτευξη ενός εναρμονισμένου επίπεδου για την προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων. Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει και ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να δώσει γρήγορα το πράσινο φως στη διαπραγμάτευση γιατί το ζήτημα επήγει για πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους. Ευχαριστώ κύριε Μπλάνκ και επιστρέφουμε στους συζητητές κύριε Χάνσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα να προσθέσω με το οποίο συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μπεγκίν ότι δηλαδή η προσχώρηση πρέπει να γίνει ήπια πρώτον και δεύτερον μετά τη σύσταση του κύριου Ντάντι ναι, οι γεωγραφικές ενδείξεις που ήδη αναγνωρίζονται από τα 7 μέλη χώρες μέλη που συμμετέχουν στη σύμβαση πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές στον κατάλογο. Αυτό, τίποτα άλλο. Και η κυρία Μπεγκίν. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Είναι αρκετά ξεκάθαρη η θέση μας. Απλώς να θυμίσω και να υπογραμμίσω ότι αν αυτό το σύστημα ήδη ίσχυε σήμερα, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε με τη Σιγκαπούρη, ας πούμε. Indeed. So... Το όντι. Τροπολογίες 21 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε με το σημείο αυτό και περνάμε στο 9. Προϋπολογισμός, μάλλον το εργαλείο για την διεθνή συνεργασία, τη γειτονία και την ανάπτυξη. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να <laughs> ε, τα συνδυάσει όλα αυτά σε ένα ε, σκέλος η κυρία Σχάκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα επικεντρωνόμαστε στη γνωμοδότησή μας για αυτό το νέο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός εργαλείου γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας, το NDICI αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για λόγου αφενή, αυτό δεν θα πρέπει να τον μπερδέψουμε με το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο ή τη γνωμοδότησή μα για το νέο ε, προταξιακό εργαλείο και τη σχετική βοήθεια. Υπάρχουν κάποιε διαφορετικέ πτυχέ ω προ τον προπολογισμό αυτών των εργαλείων. Όμω, όπω αναφέρατε και στην εισαγωγή σα με το εργαλείο αυτό, το NDICI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συγχώνευση διαφορετικών εργαλείων σε ένα. Επίση, επεξεργάζομαι το φάκελο αυτό στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και νομίζω ότι συνολικά σε ό,τι αφορά τον ε, επανασχεδιασμό του αρχιτεκτονήματο ε, των προπολογισμών για τα εργαλεία τη εξωτερική πολιτική, ένα από τα βασικά εναπομείνοντα ερωτήματα είναι πώ η νέα αυτή δομή θα ε, αποτελεί αντικείμενο χειρισμού και πώ το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει ω προ τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο. Νομίζω ότι είναι ε, προ στιγμή αδύνατο να αξιολογήσουμε τα θετικά του νέου συστήματο χωρί να δούμε τη συνολική ε, δομή και το συνολικό αρχιτεκτόνημα θα τα δουν οι συνάδελφοι ανάλογα με τις επιτροπές τις οποίες συμμετέχουν. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ευρέως ε, ανησυχίες, εμέριμνα για τη διακυβέρνηση του όλου συστήματος όπως αναφέρεται και στην έκθεσή μου ε, εκ μέρους της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Προσπαθούμε να ε, ενισχύσουμε τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της ε, εξωτερικής πολιτικής και της εμπορικής. Το έχω κάνει τονίζοντας ότι το NDICI θα πρέπει να ισχύει εμπορικές πρωτοβουλίες όπως το Aid for Trade, τους κανονισμούς ε, GSP, τη διαδικασία Kimberley και επίσης ε, τον κανονισμό για τα ορυκτά των συγκρούσεων. Επίσης το εργαλείο αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στην προώθηση και την προστασία του πολυμερού συστήματος, το οποίο δέχεται τόσες πιστέσεις, την ε, βιώσιμη οικονομική συνεργασία, τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, καθώς και τα όσα προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ. Τελευταίο, ένα από τα σημεία που ήθελα να τονίσω είναι ότι σε σχέσεις ό,τι αφορά το εμπόριο. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, συνολικά οι σχέσει μα με τι τρίτε χώρε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Περιμένω τις τροπολογίε σα με ανυπομονησία. Η προθεσμία είναι 26 Νοεμβρίου. 27. Yeah. 27, 27. Ε, το καλύτερο, λέει η κυρία Σχάκε. Ωραία, οι σκιώδεις τώρα. Παρακαλώ. Κλείνει. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ε, χαίρομαι για τη ρύθμιση αυτή που θα ενισχύσει την ευημερία, τη σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις ενδιαφερόμενες χώρες. Στην Αφρική, στις χώρες γειτονίας μας, εκεί όπου υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή θα συνεισφέρει πάρα πολύ για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές. Πρόκειται και συνεργασία με τρίτε χώρε για πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, σταθερότητα, ειρήνη, στήριξη στι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, αντιμετώπιση κρίσεων, περιπτώσεων αστάθεια, συγκρούσεων. Δίχω άλλο οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Όμως, το εργαλείο αυτό θα πρέπει να έχει και ως στόχο την ενίσχυση και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών, που είναι προϋπόθεση για μια κοινωνία που θα χαίρει σταθερότητα και ειρήνης. Οι εμπορικές συμφωνίες με επενδύσεις και καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της ρύθμισης αυτής προτείνονται μέτρα για να βοηθήσουμε και την αντιμετώπιση κρίσεων σε διάφορες χώρες. Εφόσον ε, υπάρχει ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών πολιτικών, αυτό επίσης θα βοηθήσει πολύ. Είναι διευρυμένο το πεδίο εφαρμογή με το νέο επενδυτικό πλαίσιο για τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να στηρίξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την ψηφιακή οικονομία επίσης, την απασχόληση. Θα συνεισφέρει επίσης την τοπική ανάπτυξη και θα προστατεύσει την αποστρέβλωση της ε, τοπικές αγορές. Στηρίζω λοιπόν την εισηγήτρια που λέει ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συμπληρωματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις πολιτικές μας για τις προτιμήσεις. Και τέλος, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του μέσου αυτού από το σχεδιασμό του μέχρι την αξιολόγησή του και να υπάρχει ενισχυμένος διάλογος. Αυτές λοιπόν θα είναι οι γραμμές πάνω στις οποίες θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η Γκουε, ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Σημερίζομαι εν μέρη τις ανησυχίες της για αυτό το ένα και ενιαίο μηχανισμό. Έχουμε και εμείς κάποιες ανησυχίες γύρω από αυτό το θέμα. Πρώτον, διαφοροποίηση των κονδυλίων. Κατά τη γνώμη μας ε, δεν πρέπει να ε, πέσει σε δεύτερη μοίρα η ε, διεθνής συνεργασία. Θα μπορούσε όμως, αν δεν ε, σχεδιαστεί σωστά το, ο μηχανισμός αυτός, να οδηγήσει σε τέτοιους κινδύνους για την συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης μέσω της υποταγής της διεθνούς συνεργασίας ε, γενικότερη στην γενικότερη εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Επίσης, η απουσία ε, σαφήνειας όσον αφορά τα κριτήρια ε, για την ε, υπαγωγή και τη χρηματοδότηση από το μηχανισμό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τα παραδοτέα, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ανθρώπινοι δικαιώματα θα, πρέπει να, θα έπρεπε να αποτελούν το βασικό κριτήριο των, ε, της χρηματοδότησης. Οι πόροι που θα κατανέμονται πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν αν δεν ε, γίνουν σεβαστά αυτά τα κριτήρια. Για τους δικαιούχους, ο ένας και νέος μηχανισμός σημαίνει ότι ε, κάποια συμμετρικά προγράμματα θα χαθούν. Αυτό έχει προκύψει και από την εμπειρία μας. Η ενιαία αυτή στάση λοιπόν και ο νέος μηχανισμός μπορεί να πλήξει ορισμένες περιοχές, περιφέρειες ε, ή και ορισμένους τομείς πολιτικής όπως είναι η ισότητα των φίλων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής βοήθειας να ε, κατευθυνθεί στις χώρες LDC. Σήμερα στις ε, ε, περισσότερες ε, χώρες ε, ε, ε, πρέπει να σεβαστούν τον στόχο του 0,2% του ΑΕΠ. Για τη δημοκρατική συμμετοχή εμείς θέλουμε να υπάρχει πλήρης δημοκρατική, δημοκρατικός έλεγχος και συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση. Και πέμπτον, η ευελιξία ε, ε, θυσιάζεται ε, υπέρ της ε, αποτελεσματικότητας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια προσέγγιση που μπορεί να ενισχύσει τους κινδύνους ε, και να θέσει σε κίνδυνο το, την μακροχρόνια στόχευση του μηχανισμού. Τέλος, το είχα πει και γενικά για το πι δέλτα πι, είμαστε ανήσυχοι γύρω από αυτήν την προσέγγιση για τον ενιαίο μηχανισμό εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για άλλη μια φορά και σε αυτή την κατεύθυνση θα συζητήσουμε με, τους, με την εισηγητρία. Κυρία Χάουταλα για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια ε, εισηγήτρια η οποία γνωρίζει το αντικείμενο καθώς ε, χειρίζεται τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή Εξωτερικών Επιθέσεων. Κάτι γενικό πρώτα. Η ομάδα μου συμφωνεί ότι χρειάζεται απλούστευση και συμπράξεις μεταξύ των 12 μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης. Έχουμε όμως κάποιες αμφιβολίες ε, οι οποίες δεν αφορούν τόσο την Επιτροπή Ίντα. Γενικά πιστεύουμε ότι ε, θα μπορούσαν να συγχωνευτούν έξι μηχανισμοί ε, εξωτερικής χρηματοδότησης και πέντε μέσα ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά κάποια, θεωρούμε, κάποια μέσα θεωρούμε ότι θα έπρεπε να παραμείνουν ξεχωριστά. Υπάρχουν ανησυχίε εδώ στο Κοινοβούλιο για την συγχώνευση όλων αυτών των μηχανισμών σε έναν μηχανισμό. Αν όμω γίνει τελικά αυτή η συγχώνευση θα πρέπει να συνοδεύεται από εχέγγυα και η συγγήτρια νομίζω ότι καλώ επεσήμανε τη σημασία τη διακυβέρνηση αυτού του μηχανισμού. Να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπωσδήποτε στον έλεγχο των πεπραγμένων αυτού του μηχανισμού. Επίσης, εκτιμώ τις τροπολογίες της εισηγήτριας που τονίζουν τη σημασία των μηχανισμών εμπορίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Τροπολογία 3, 7 ε, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των ε, παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Γιατί αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της εξέτασης του πώς μπορεί το εμπόριο να ωφελήσει και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα ήθελα να υποβάλω και εγώ μια τροπολογία. Να υπενθυμίσουμε δηλαδή στην Κομισιόν ακόμη περισσότερο την ανάγκη να θεσπίσει ε, την δέουσα επιμέλεια οριζοντίως. Έχουμε εξαιρετική νομοθεσία η οποία αναφέρεται στην τροπολογία 3 τη διαδικασία Κίμπερλι, έχουμε την, τον κανονισμό για, τις, ε, ο, για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Θέλω να υπενθυμίσω και τον κανονισμό για την ξυλία που έχουμε, που επίσης είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ε, το οποίο πρέπει να ε, γίνει σεβαστό στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξία. Νομίζω ότι το σχέδιο κειμένου που έχουμε μπροστά μα είναι εξαιρετικό. Κάποιε τροπολογίε θα υποβάλω εγώ, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση που μόλι περιέγραψα. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου τη ΙΝΜΑ, τη σκιώδου ε, εισηγήτρια του Σοσιαλιστή, θα σα πω εγώ τη θέση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δυστυχώ η ΙΜΑ ε, δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα στην Επιτροπή μα. Καταρχά, χαιρετίζει το σχέδιο κειμένου τη κυρία Σχάκε και έχει κάνει κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις. Οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν τη συγχώνευση των, μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης και ιδίως τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που αποτέλεσε ε, μακροχρόνιο αίτημα τόσο του Κοινοβουλίου όσο και των Σοσιαλιστών. Ο προτινόμενος προϋπολογισμός των 89,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θεωρούμε ότι θα εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, ε, πολιτικών εμπορίου και ε, ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βιωσιμή ανάπτυξη. Επίσης, σημαντική είναι η υπεράσπιση του πολυμερού συστήματος εμπορίου με τον ΠΟΕ στο επίκεντρό του. Γι' αυτό χρειάζεται μηχανισμός χρηματοδότησης για την υποστήριξη του εξοχρονισμού του ΠΟΕ για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογής των ε, συμφωνιών εμπορικής διευκόλυνσης αλλά και για την επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ του ΠΟΕ και άλλων διεθνών οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είναι ο ΆΕΛΟ, η UNCTAD και η UN Women το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της ε, διαφάνειας και της λογοδοσίας. Από αυτή την άποψη χαιρετίζουμε την αναφορά της εισηγήτριας στην ανάγκη ε, ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη δημοσιονομική διαδικασία. Επίσης, χαιρετίζουμε την αναφορά στη σημασία εξασφάλισης ορθής εφαρμογής του μηχανισμού Aid for Trade για την δέουσα επιμέλεια, για τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες και τον κανονισμό ε, για την καταπολέμηση των βασανιστήριων, τη διαδικασία Κίμπερλι και τον κανονισμό GSP. Η ίνμα θα ήθελε επίσης να γίνονται και κάποιες άλλες ρητές αναφορές στο κείμενο, όπως στην ανάγκη να βελτιωθεί η εξάντε και εξπόστα αξιολόγηση των ε, ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, την ανάγκη να γίνουν τα κεφάλαια για το εμπόριο πλήρως εκτελεστά με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχουν οι συμφωνίες και τη σημασία της παροχής τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας στους εμπορικούς μας εταίρους προκειμένου να μπορούν να συμμορφώνονται με τα δικά μας πρότυπα. Η ΕΜΑ λοιπόν προσβλέπει σε μια καλή συνεργασία επικοδομητική με την εισηγήτρια. Δεν ζήτησε κάποιος άλλος το λόγο. Οπότε θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράτης από την Κομισιόν ο κύριος Δημητρίου από την DG DEFCO. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τις τροπολογίες της κυρίας Χάκε που υπογραμμίζει την μνήα του Trade for Aid. Πράγματι, το εμπόριο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπέρ αξιών και αρχών. Το εμπόριο συμπεριλαμβάνεται ήδη στον κανονισμό, στο άρθρο 3, 5, τις συνθήκες όπου το εμπόριο είναι ένας από τους στόχους. Αναφέρεται λοιπόν και στο, στη ρύθμιση ως ένας από τους κύριους στόχους, όπως επίσης και στους στόχους του 2030 και την Ευρωπαϊκή Συνένεση. Οπότε η όθηση του εμπορίου είναι ένας από τους κύριους στόχους της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Και όπως και εσείς και εμείς πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν από τον μηχανισμό για να δημιουργηθούν επενδύσεις, να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση δημιουργώντας ε, οδούς μετανάστευσης κτλ. Εμείς, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, θέλουμε ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην ΑΦΕΤ. Και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει, να δίνει πολιτική κατεύθυνση στην υλοποίηση αυτού του εργαλείου. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο είναι για την αναπτυξιακή βοήθεια. 92% του συνολικού ποσού του μηχανισμού πηγαίνει στην ανάπτυξη και έτσι πρέπει να καταγράφεται ως αναπτυξιακό μέσο. Είναι η μεγαλύτερη συνιστόσα του μηχανισμού αυτού η ανάπτυξη. Άκουσα ε, για αυτά που είπατε για την ελαστικότητα σε σχέση με την ε, προβλεψιμότητα. Και στο αναπτυξιακό ταμείο, κάτι που έχει ζητήσει εδώ και καιρό το Κοινοβούλιο, προτείνουμε ένα ποσό το οποίο δεν διατίθεται συγκεκριμένα σε κάτι. Δεν είναι με 20%, είναι περίπου 11%. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και κάποια κατεύθυνση για αυτό το ποσό. Πάντως, χωρίς το αναπτυξιακό ταμείο που έχει 20% δεν θα ήμασταν σε θέση να αντιμετωπίσουμε αλλαγές που προκύπτουν, όπως ήταν το έμπολο, για παράδειγμα, όπως ήταν η μεταναστευτική κρίση. Για το EFSD, για το Ταμείο Επενδύσεων, το Juncker, όπως το λέμε, η ο νέος αυτός μηχανισμός χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και εκεί. Υπό τον χρηματοδοτικό κανονισμό, όσον αφορά δηλαδή τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Ανάπτυξης ΣΥΝ, έχουμε πλήρη εφαρμογή των όσων αναφέρονταν πριν και εδώ. Προσβλέπουμε στην τελική γνωμοδότηση, στις τροπολογίες και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να χτίσουμε με το μηχανισμό αυτό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στην εξωτερική δράση μέσω ενός μηχανισμού. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα σας. Και εμείς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ικανοποιημένοι από, ε, από το κείμενο και τις τροπολογίες της Επιτροπής σας, γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνουν και το πνεύμα της δημιουργίας ενός μηχανισμού για την εξωτερική συνεργασία που να καλύπτει ε, βρέως διάφορες πολιτικές για την ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν και με το εμπόριο, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, μας ικανοποιεί τα όσα αναφέρονται για την εμπορική πολιτική, για την οικονομική διπλωματία, για μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την απασχόληση και όλος ιδιαίτερος μας ικανοποιεί το ότι υπογραμμίζεται η πολυμερής διάσταση. Κάτι πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε λοιπόν την διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή σας. Για το θέμα της διακυβέρνησης του μηχανισμού. Όπως προτείνεται, είμαστε υπέρ της συνεχούς ενημέρωσης όσον αφορά την υλοποίηση του μηχανισμού Θέλουμε να έχουμε τακτικά ανταλλαγή απόψεων με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και επίσης, να ξέρετε ότι μας αρέσει η πρακτική της Επιτροπής σας που έχει μία ομάδα ελέγχου για τις εμπορικές συμφωνίες. Οπότε και από αυτού θα φροντίσουμε να έχουμε τακτικά επαφές. Είναι πολύ πολύ ο έλεγχος του Κοινοβουλίου ακόμη και σε καθημερινή βάση. Θέλω επίσης να σας πω ότι συμφωνώ με διάφορα σχόλια που ακούστηκαν από την κυρία Χαουτάλα, για παράδειγμα, η οποία είπε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια των αλυσίδων προμήθειας. Συμφωνώ και εγώ με αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Επίσης, ανθρώπινα δικαιώματα, διαφάνεια στη λογοδοσία, και προδιαγραφές περιβαλλοντικές προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικά στο δικό μας έργο. Και βέβαια η στήριξη των επενδύσεων που έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Οπότε περιμένουμε και εμείς να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποφασίσει η Επιτροπή σας. Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Σχάκερ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει εδώ μεγάλο περιθώριο να καταλήξουμε σε μία ε, γνωμοδότηση με βρία συνένεση. Και εγώ, μετά από αυτά που άκουσα από την Επιτροπή, και εγώ θα ήθελα να ξέρω πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα το ότι συμβαίνει. Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις είχαμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα περί διακυβέρνησης πριν αξιολογήσουμε το μηχανισμό. Οπότε πρέπει να θέσουμε τις προτερότητές μας και είναι να μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε όλη την πορεία ότι υπάρχει καλή διακυβέρνηση και τα κονδύλια δαπανώνται σωστά. Βλέπω ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οπότε ελπίζω ότι θα αντικατοπτρίζεται και στο κείμενο αυτό που είπαν και συμφωνώ και εγώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. 27 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στις 6 μετά μεσημβρίας. Ωραία, φτάνουμε στο σημείο 10 που είναι ε, η αντιπροσωπεία του hoc που πήγε στο κοινοβουλευτικό φόρουμ G20 στο Μπένος Άιρες. Παρακαλώ, ο επικεφαλής να μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Μια αντιπροσωπεία εννέα μελών επισκέφθηκε τον Buenos Aires ε, και το κοινοβουλευτικό φόρουμ του G20. Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων εκπροσωπήθηκαν και επίσης μας συνόδευσαν τέσσερις συνεργάτες της Επιτροπής μας. Η συνολική μου εικόνα είναι θετική. Ήταν επιτυχής η επίσκεψη και από άποψη επιμελητίας και διοργάνωσης πολύ περίπλοκη. Ήταν το πρώτο κοινοβουλευτικό φόρουμ στο επίπεδο του G20 και ήταν το πρώτο διότι όλες οι άλλες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν είχαν οργανωθεί στο παρελθόν σε διαφορετικό επίπεδο και όχι με τόσο καλή εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων των μέλων του G20. Ο κύριος Μακάλιστερ και εγώ ο ίδιος συμμετείχαμε σε, πολλές, σε πολλά πάνελ συζήτησης για την αποτελεσματική και διαφανή διακυβέρνηση χωρίς διαφθορά με τη συμμετοχή του Προέδρου κύριο Μακάλιστερ και το βιώσιμο εμπόριο για μένα από την Ίντα. Είχαμε πολλές ανταλλαγές απόψεων σε πολυμερές επίπεδο και περιφερειακό με εκπροσώπους κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών και πριν και μετά το κοινοβουλευτικό φόρουμ. Ήταν σημαντική στιγμή αυτή της επισκέψής μας για τις σχέσεις με τη Μαρκοσούρ και τη Συμφωνία Σύνδεσης που μπορεί να συνεχθεί και αποστήλαμε ένα ηχηρό μήνυμα στήριξη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μα, πριν τι ευρωεκλογέ. Βεβαίω, μιλάμε για μία περίοδο λίγο μετά τι προεδρικέ εκλογέ στη Βραζιλία και αυτό ήδη έχει αρχίσει να αφήνει τον αποϊχό του και τον αντίκτυπό του στις τάσεις και το τι κατεύθυνση μπορεί να πάρουν οι με τη Μαρκοσούρ. Ε, συζητήσαμε ομάδες φίλων από την ε, γερουσία της Αργεντινής, είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον από αυτούς και αν έπρεπε να σταθώ σε ένα αρνητικό τη αποστολή, θα έλεγα από το επίπεδο κάποιων των συναντήσεων. Περιμέναμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο τη Αργεντινή, αλλά δεν ήταν δυνατό αυτό. Και μια-δυο συναντήσει τελικά υποβαθμίστηκαν ως προς το κλιμάκιο των ε, συνομιλητών μας. Από υπουργό πήγαμε σε υφυπουργό ή εκπρόσωπο του Υπουργείου και ούτω καθεξής. Δύο πράγματα ακόμη θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα ότι απειλείται η κοινοπολιτική διάσταση του G20. Είναι σημαντικό ήδη φέτος ε, να επαναλάβουμε αυτό που έγινε στον Πένος Άιρες και να είμαστε πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια για τις συναντήσεις του G20. Και το δεύτερο είναι η παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ που είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα συμπεράσματα. Έχω χρόνο νομίζω, Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα η δημιουργία του κοινοβουλευτικού φόρουμ του G20 νομίζω ότι είναι σαφές να το καλωσορίσουμε. Όλοι μας οι συνάδελφοι, οι βουλευτές των χωρών G20 καλωσόρισαν την πρωτοβουλία αυτή διότι αυξάνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας G20. Μέχρι τώρα είχαμε τις συνόδους των ηγετών, των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα έχουμε το κυβερνητικό φόρουμ να το διατηρήσουμε. Μετά για τη χώρα υποδοχή στην Αργεντινή, νομίζω ότι όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας είδαν ότι το άνοιγμα της Αργεντινής μετά από δεκαετίες απομόνωσης ε, και προστατευτισμού είναι ε, πραγματικότητα. Έχουν δεσμευτεί ω προ τη διεθνή συνεργασία, την πολυμερή προσέγγιση και το ελεύθερο εμπόριο. Βεβαίω υπάρχει ανάγκη οι προσπάθειέ του να ενταθούν. Πρέπει και αυτοί από την πλευρά του να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών και διαφορετικών ομάδων του πολιτισμού στην όλη προσπάθεια για τι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ ε, δείξαμε την ε, ξεκάθαρη στήριξή μας και σε επίπεδο δηλώσεων τα είπαμε και στην έναρξη της, ε, του φόρουμ, αλλά ξέρουμε τώρα ότι είναι ο νέος πρόεδρος ο κ. Μπολσονάρο στη Βραζιλία, οπότε η κατάσταση δεν θα είναι εύκολη. Η περιφερειακή κατάσταση, οι σχέσεις μεταξύ των μελών του Μερκοσούρ δεν είναι εύκολη. Επίσης, επειδή έχουμε... Είχαμε συνάντηση βουλευτών από τόσο διαφορετικέ χώρε. Μπορέσαμε να εκφράσουμε και προτάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο επίπεδο του ΠΟΕ. Η ανάγκη μεταρρύθμισης που παγκοσμίως αναγνωρίζεται ε, θα πρέπει να προχωρήσει. Βεβαίω τώρα το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης και τη ανανέωση είναι κάτι που δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί. Και για να ολοκληρώσω, η συνεργασία ε, των ε, φορέων και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε πολύ καλή στήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Buenos Aires ε, με την ε, συνδρομή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Είχαμε γραπτή απενημέρωση από την ΙΕΤ. Βέβαια πρέπει να πω, και συγγνώμη που θα ολοκληρώσω με αυτό, ότι ζητήσαμε και η ΑΦΕΤ και η ΙΝΤΑ ε, απενημέρωση από την ε, DigiTrade, το οποίο δεν λάβαμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Αλλά συνολικά ήταν πολύ καλή η επίσκεψή μας και ελπίζω ότι νομίζω ότι μάλλον ότι πετύχαμε να επιδείξουμε ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των ε, συναδέλφων διαφορετικών πολιτικών ομάδων, προκειμένου να περάσουν τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κοινοβουλευτικές μας αξίες και το ενδιαφέρον μας για το μέλλον. Νομίζω ότι αφήσαμε το σημάδι μας αυτή την εκδήλωση του G20 και γραπτός αλλά και με τα οπτικό ε, το οπτικοακουστικό υλικό που ε, έμεινε από τον Πένος Τέλεια. Ερωτήσεις, σχόλια, κύριε Σόλτς. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον επικεφαλής για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Ίσως δεν άκουσα καλά. Αλλά έπαιξε κάποιο ρόλο το φόρουμ για το Χάλιβα στο G20. Διότι το G20 έχει υπό την Κινέζικη Προεδρία συστήσει ένα φόρουμ για το Χάλιβα και όποτε ρωτάμε, ζητάμε την εξέβρεση λύσεων και από την DG εμπορίου, υπενθυμίζουμε ότι και αυτό το φόρουμ για το χάλιβα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν ξέρω λοιπόν, θα ήθελα να, να μου πείτε αν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στο Buenos Aires. Δεύτερο ερώτημα. Είπατε για τις συζητήσεις που είχατε για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Υπάρχει κάποια ευαισθητοποίηση ιδίως από τους εκπροσώπους των πιο ανεπτυγμένων χωρών του Νότου για να συνδεθούν τα εμπορικά ζητήματα με τα ζητήματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. ερώτηση. Εκπροσωπήθηκαν και τα 20 ε, μέλη του G20 στην κοινοβουλευτική διάσκεψη και ποια ήταν η συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών των κοινοβουλευτικών των διαφορών χωρών. Okay, thank you very much. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι δεν συμμετείχε η Αμερικανική αντιπροσωπεία, δεν υπήρχαν μέλη του Κογκρέσου δηλαδή στην κοινοβουλευτική αυτή διάσκεψη. Γι' αυτό και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας πώς ήταν η συνεργασία μας μαζί σας. Βεβαίως ήταν αντικείμενο συζητήσεων η ΕΠΑ. Αυτό είναι σαφές αλλά δεν είναι το ίδιο. Συζητήσαμε επίσης και κατά τη διάρκεια των πάνελ. Υπήρξαν λοιπόν κάποια πάνελ με αυτή ήταν η μορφή των συζητήσεων που ακολουθήθηκε και στη συνέχεια ε, υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων μετά τις παρουσιάσεις των ομιλητών και εκεί συζητήθηκαν εκτενώς οι θέσεις των ΙΠΑ και οι πιθανές εξελίξεις ε, που θα προκύψουν από διάφορες αποφάσεις που λαμβάνει ο πρόεδρος των ΙΠΑ γύρω από δασμολογικά θέματα και επίσης εκφράστηκε και μια κάποια δυσπιστία απέναντι στη ΣΥΠΑ στο πλαίσιο ε, του ΠΟΕ. Εκείνοι που τουλάχιστον τοποθετήθηκαν στην κοινοβουλευτική διάσκεψη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον ΠΟΕ, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού αυτού. Δεν μιλήσαμε για την ουσία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν, ε, οι συμμετέχοντες συζητήσεις δεν είχαν αυτό το επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για να εισέλθουν σε λεπτομερή συζήτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όλα αυτά χωρίς παρουσία των ΗΠΑ. Για το φόρουμ, για το χάλιβα, η απάντηση είναι παρόμοια, κύριε Σόλτς. Το G20 στη σύνοδο κορυφής του στην 1η Δεκεμβρίου θα συζητήσει αυτό το θέμα. Εμείς το θέτουμε βεβαίως το φόρμα αυτό. Εγώ συμμετείχα και σε ένα πάνελ για την πολυμέρεια και εκεί ε, ε, ένας εκπρόσωπος της Κορέας έθεσε το ζήτημα της ε, υπερπαραγωγής χάλιβα. Σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη τώρα, Χέλμουτ, νομίζω ότι ήταν ε, το πλέον εμφανές και ορατό θέμα που απασχόλησε τις συζητήσεις μας. Πολλοί άριθμοι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, στους στόχους για το 2030 και επισήμαναν την ε, ανάγκη σε όλες τις νέες εμπορικές πολιτικές να ε, συμπεριλαμβάνεται αυτή η διάσταση. Να σας πω επίσης ότι κάποιοι αναλυτές όχι οι συμμετέχοντες ε, στην διάσκεψη, αλλά σε επίπεδο αναλυτών, εκφράζεται ε, ένας σκεπτικισμός, ε, μια επιφυλακτικότητα απέναντι στον, στην κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη, με το επιχείρημα ότι η εκτελεστική εξουσία βεβαίως εναπόκειται στις κυβερνήσεις. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά σημαντικό για μας είναι να επιβεβαιώσουμε τον, τον ρόλο μας ως ε, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Για τις είπα να σας υπενθυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι είχαμε τις ενδιάσιμες ε, εκλογές στην περίοδο που έγινε η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη του G20 και ίσως γι' αυτό απήχαν ε, οι γερουσιαστές των ΗΠΑ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε το σημείο 10 και περνάμε στο 11, πρώτη ψηφοφορία. Έχουμε ένα λεπτό μέχρι να ξεκινήσουμε. Α, κύριε Χάντζεν, με συγχωρείτε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάτι το οποίο ήθελα να θέσω, διότι η γραμματεία της ΣΥΝΤΑ μας ενημέρωσε ότι αποστήλατε επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, στην Άμπε, εξ ονόματος των Πρόεδρων και Αντιπροέδρων της ΙΝΤΑ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιστολή με εξέπληξε διότι δεν διαβουλευτήκατε μαζί μας για το θέμα αυτό. Συζήτησα και με άλλους και συζητητές. Δεν είχε προηγηθεί συζήτηση, ούτε αποφασίσαμε σε επίπεδο Επιτροπής ΙΝΤΑ. Οπότε πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος ασέδωσε έδωσε ε, την εντολή να αποστείλετε τέτοια επιστολή. Επίσης, το βρίσκω αρκετά περίεργο που αποστήλατε την επιστολή αυτή απευθείας στον κύριο Άμπε, διότι κανονικά θα έπρεπε να αποσταλεί απευθεία στην αντιπροσωπεία μας εδώ, ε, την αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε μάλιστα στα πρώτο πληθυντικό στην επιστολή αυτή, λες και πρόκειται για όλους μας εδώ, γιατί δεν ξέρω αν μιλή, ε, εκφραστήκατε προσωπικά ή εκ μέρους όλης της Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι εκφράσατε απόψεις όλων και είπατε ότι θέλετε να έχετε νέα στοιχεία για το κεφάλαιο TSD πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, μάλλον στην Ολομέλεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποια είναι η στρατηγική σας με αυτό το αίτημα. Διότι είχαμε συνάντηση της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας ε, στο Στρασβούργο και ο εισηγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μα είπε ξεκάθαρα τι έγινε στι συναντήσει που έχουν ε, μεσολαβήσει. Θα ήταν καλό λοιπόν να ενημερώνεστε και από τον εισηγητή ε, που είναι, που με το θέμα αυτό. Πραγματικά λοιπόν ε, ευνηδιάστηκα πάρα πολύ και έχω τρομερές, τρομερές για το περιεχόμενο της επιστολής αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρατηρήσεις. Πράγματι, εγκρίναμε ένα ψήφισμα εδώ στην Επιτροπή μας και θεωρήσα ότι είναι καθήκον μου να ε, πω στους Ιάπωνες ότι υπάρχει πλειοψηφία στην Επιτροπή μας υπέρ της συμφωνίας. Πού είναι ο στόχος. Και ανέφερα κάποια σημεία ε, που συζητήθηκαν ε, και στο ψήφισμα. Το, τα είπαμε χθε και με τους συντονιστές αυτά. Και καταλήξαμε ότι προτού ξανααποσταλεί τέτοια επιστολή θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και με τους συντονιστές. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία. Not working. So, everybody has Ψηφίσατε όλοι. Το δοκιμαστικό. Τέλος. Όλα φαίνεται ότι λειτουργήσαν καλά. Οπότε. Είμαι υπέρ. Αν είναι η πραγματική ψηφοφορία. Εγώ νόμιζα ότι κάνατε δοκιμαστική ψηφοφορία. Δεν παρακολούθησα. Όχι, δοκιμαστικό ήτανε. Δοκιμαστικό ήτανε. Ωραία, υπερψηφίζω. Τώρα περνάμε στην πραγματική ψηφοφορία και ψηφίζουμε την τεχνολογία blockchain της Emma McClarkin. Πρώτη τροπολογία είναι συμβαστική τροπολογία αριθμός 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Ξέχασα την 31 του Κλάου Μπούχνερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε 63. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. 64 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω το απορρευτικέ, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 95. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ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 Απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε καλού κακού. Για την 6 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Τώρα. Γνωμοδότηση Ήτρε. Πρέπει να ψηφίσουμε την παράγραφο 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Μακλάρκιν. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 12. Είναι η... Ο εξυγχρονισμός του ΠΟΕ είναι θέμα που το έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες επί μακρόν και με διάφορες αφορμές. 10, 12, 12. 12. Yeah. Wrong list or wrong number. was there a change of agenda, ah, Okay, so to be clear, it's item 12. Λοιπόν, Ξαναλέω. Σημείο 12. ΠΟΕ. Εγώ και ο κύριο Ρούμπικ είμαστε συνεισηγητέ. Πρώτα, ε, συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και επιπλέον προς την ε, ε, συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προσθήκη δηλαδή. 43. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη προς την ε, συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ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 4, σας παρακαλώ. Γιατί δεν καλύπτεται από την ε, συμβαστική 31. Η γραμματεία λέει ότι αυτό δεν συνάδει με την συμβαστική τροπολογία. Τι λέτε κύριε Ρούμπιχ, εσείς τι πιστεύετε. Ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν επί της παραγράφου 4 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και Περνάμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. And the vote is... Πέρασε. Ωραία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Πλέον έχουμε θέση για, την, για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Επόμενο θέμα, το σημείο 13 προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης. Έχουμε τροπολογία 1. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ε, εξηγήσω κάτι, διότι υπήρξε μια συζήτηση για το παραδεκτό. Εφόσον η Σαμόα είναι στις, στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τον μηχανισμό πίεσης που έχουμε. Γι' αυτό και προτείνω το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. Σημείο 14. Ετήσια έκθεση 2017 σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ κατά αποχές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 Α ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ επί τη συμβαστική τροπολογίας 3. Πέρας. Ναι, όχι. Σαφώς απερίφθη. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Όχι, καταπίπτει, συγγνώμη, καταπίπτει 19. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Με αποχέ απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε θέλετε, παρακαλώ, βεβαίω. Άρχεται η ψηφοφορία επί τη τροπολογία 24. Πέρα. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 32. Πέρας. Τώρα ξαφνικά είναι όλοι υπέρ, Ε, ε όχι και όλοι, αλλά πάντως εγκρίνεται. 35 και 36, 37 που ταυτίζονται υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές. Ψηφίζουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Τώρα, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Α, εγκρίνεται. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι σίγουρο, οπότε καλύτερα να το επαληθεύσουμε μέσω ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ επί του συνόλου του σχέδιου γνωμοδότηση. όπως τροποποιήθηκε. And the vote ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ισηγητά Και με αυτό ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία και περνάμε στο σημείο 15. Αν κάποιος θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, αλλά σας παρακαλώ ησύχως. 15. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Έγινε μια ομάδα παρακολούθηση για το GSP. Θέλω να δώσω το λόγο στον Κρίστοφ Γένερτ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. 16 Οκτωβρίου είχαμε μια ομάδα ελέγχου για το ΕΣΠΗ και επικεντρωθήκαμε σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα την άρση του ε, όλεκτος από όπλα με την ε, Καμπότζα και μετά συζητήσαμε και την ε, μεσοπρόθεσμη έκθεση. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για την ερευνητική αποστολή στην Μιαμάρα και για το ότι δημοσιεύθηκε η άρση στην επίσημη εφημερίδα. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει ένα χρόνο και μπορεί να καταλήξει είτε σε μία άρση, σε πλήρη άρση, σε μερική άρση. Όλες οι εναλλακτικέ δηλαδή υπάρχουν. Υπογραμμίσαμε πόσο σημασία έχει οποιαδήποτε άρση να λάβει υπόψη το συνολικό στόχο του SP και δηλαδή και την ανακούφιση από τη φτώχεια, την βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. Γιατί πιστεύω, ξέρουμε ότι είναι σοβαρή η κατάσταση στην Μιαμάρ και στην Καμπότζα, αλλά υπάρχουν θέματα σημαντικά όπως είναι απασχόληση για τις γυναίκες και άλλοι παράγοντες εδώ που διακυρδεύονται και δεν θα έπρεπε να απειληθούν από αυτό που θα κάνουμε. Η Επιτροπή επίσης μας ενημέρωσε για την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του προγράμματος και σημείωσαν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για τη μελέτη δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για ολόκληρη την τετραετία που εμείς αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτά έχω να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις για το GSP. Όχι από ό,τι βλέπω. Επόμενη ομάδα ελέγχου. Ηνωμένε Πολιτείε με Καναδά και Μεξικό. Αυτή είναι η επόμενη ομάδα. Συζητήσαμε εδώ βέβαια για την ΑΦΤΑ. 2-0, τώρα ονομάζεται UMCA. Στην ναι, αυτή συμφωνία ναύτα υπάρχουν κάποιες διατάξεις που κατά τη γνώμη μας δεν ευθυγραμμίζονται με τον ΠΟΕ. Για παράδειγμα η διπλή προέλευση ποσοστά προϊόντων, ότι ένα ποσοστό πρέπει να παράγεται σε μια χώρα που να έχει τουλάχιστον 60 δολάρια. Και επίσης για το Μεξικό, ποσοστώσεις εξαγωγών που πρέπει να γίνονται αποδεκτές και η απειλή για τους δασμούς επίσης υπάρχει στη συμφωνία. Συζητήσαμε τη συμφωνία λοιπόν και στείλαμε καθαρό μήνυμα στην Επιτροπή ότι θέλουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς και κατασκευαστές και μας υποσχέθηκαν ότι θα τα έχουμε σύντομα. Αυτά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ο εισηγητής μας για τον Καναδά, ο κύριος Παύλης, έφυγε από το Κοινοβούλιο και δεν έχουμε αντικαταστάτη. Το ΕΛΚ νομίζω ότι πρέπει να δώσει κάποιο όνομα. Ωραία. Καλώς. Ερωτήσεις. Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Και πάμε στην ad hoc αντιπροσωπεία στη Νότια Αφρική. Η κυρία Σχάκια ήταν και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Πήγαμε στην Νότια Αφρική 29 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου. Οποιοςδήποτε παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτή τη σημαντική χώρα της Αφρικανικής Επίρου γνωρίζει ότι υπάρχει μια μεγάλη μετάβαση στη χώρα μετά την κυβέρνηση Ζούμα. Τώρα έχουμε τον πρόεδρο Μαπόζα, ο οποίος ήρθε μάλιστα στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και μας παρουσίασε τις απόψεις του μετά από την επίσκεψή μας εκεί. Η επίσκεψη αυτή ήταν μια ευκαιρία για να καταλάβουμε καλύτερα για αυτές τις αλλαγές στη Νότια Αφρική και να επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Μπόρντο, ο οποίος μας εξήγησε πώς προσπαθεί η νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και όλη την προβληματική στην Νότια Αφρική με τις μεταρρυθμίσεις των κρατικών ε, επιχειρήσεων και πώς θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να μιλήσουμε με επιχειρηματίες γυναίκες για το πώς ε, μπορούν ε, να βοηθηθούν μέσω του εμπορίου. Συζητήσαμε και πολύ καλά για τη γεωργία, για εντάσεις που δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Αφρική, αλλά ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια διέξοδος εκεί. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ένα ορυχείο ε, πλατίνας, όπου έτσι καταλάβαμε και το εύρος, δηλαδή πόσο μεγάλο είναι αυτό το ορυχείο, τι επιπτώσεις έχουν τα έργα αυτά στις τοπικές κοινότητες, με τις οποίες μιλήσαμε, με εκπροσώπους τους δηλαδή, μετά την επίσκεψή μας στο Ρηχείο. Επίσης, μάθαμε και για τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατανομή της γης, γιατί μετά το Apartheid δεν υπήρξε αύξηση της ιδιοκτησίας γης από τους μαύρους. Οπότε οι εντάσεις, όπως καταλαβαίνετε, παραμένουν. Και βέβαια είναι δύσκολη λύση, γιατί Υπάρχουν αγρότες που έχουν μεγάλη διοκτησία και δεν θέλουν να παραιτηθούν από αυτή, ακόμα και αν πολλοί υποστηρίζουν την ανακατανομή για να υπάρξει καλύτερη ισορροπία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Επίσης πήγαμε στο Cape Town από το Johannesburg και είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ε, αμπέλια που λειτουργούν με προοδευτικό τρόπο, δηλαδή εκπαιδεύουν παιδιά από διαφορετικά υπόβαθρα, επιτόπου, πιστεύουν πολύ στην εκπαίδευση και επιστρέφουν, επιστρέπουν και spin-offs, δηλαδή νέα μπέλια από αυτούς οι οποίοι δούλευαν παλιά στις μεγάλες ε, καλλιέργειες και τώρα αυτοί φτιάχνουν κάποιες μικρές καλλιέργειες και φτιάχνουν το δικό τους κρασί. Τους βοηθούν. Είναι από τις καλύτερες πρακτικές. Άρα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συναντηθούμε με όλους αυτούς, να μάθουμε περισσότερα για τις αλλαγές αυτές που λαμβάνουν χώρα στη Νότια Αφρική. Και ελπίζω ειλικρινά ότι και εμείς πήγαμε εκεί και ο πρόεδρος τους ήρθε εδώ. Αυτό θα ενισχύσει τις σχέσεις μας ε, μαζί τους. Σίγουρα ε, η ε, Νότια Αφρική βλέπει τον BRICS μια νέα δυνατότητα έτσι, ολοκλήρωσης με πολλές ελπίδες, αλλά θα δούμε πού θα καταλήξει. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι παρά το δύσκολο παρελθόν και πρέπει και εμείς να είμαστε τα πινόφρονες, να ξέρετε ότι τώρα προχωρούν με μέτρα από τα οποία αποφελεί το κόσμος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Είναι όντως περίπλοκη η κατάσταση στην Νότια Αφρική με πολλές αλλαγές. Και δικιά μου αίσθηση είναι ότι οι σχέσεις της Νότιας Αφρικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από διάφορα πάνω και κάτω. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας μας, η οποία περιέγραψε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ε, Νότια Αφρική, αλλά και γενικότερα την κατάσταση στην περιοχή. Οι εξαγωγές προϊόντων ποιότητας συνεισφέρουν οι διάφορες ομάδες πληθυσμού να έχουν μια προσέγγιση μεταξύ τους για τα θέματα της εκπαίδευσης. Εγώ είδα τα σχολεία τα οποία δημιουργήθηκαν στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσα. Ήταν θεματικό δείχνει ότι η αγροτική μεταρρύθμιση στη Νότια Αφρική έχει τις προϋποθέσεις και για περισσότερη παραγωγικότητα. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις, ιδιοκτησίες και το κράτος πρέπει φυσικά να βρει τον τρόπο να αποδώσει σε ιδιώτες γη. Τότε θα είναι χρήσιμη αυτή η μεταρρύθμιση. Όταν πήγαμε στο ρηχείο, εξεπλάγει πάρα πολύ. Υπήρχε και κοβάλτιο που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. 7 κιλά κοβάλτιο χρειάζονται ανά μπαταρία. Επί 3 πολλαπλασιάζουμε για την τιμή, η οποία όμως δεν καλύπτει ακόμα. Άρα εδώ πρέπει να γίνουν πράγματα για τις πρώτες ύλε. Και βέβαια αναρωτηθήκαμε πώς ανακυκλώνεται μετά το κομπάλτιο. Γιατί δεν πρέπει να το πετάμε απλώς και να βρούμε και τρόπους ανάκτησης του κοβαλτίου από τις μπαταρίες. Οι συζητήσεις ήταν πολύ έντονες και πολύ ενδιαφέρουσες πώς δηλαδή σε μια κυκλική οικονομία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Εγώ τουλάχιστον έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όλοι μάθαμε πολλά εκεί. Ήταν για όλους μας πάρα πολύ χρήσιμο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τη Μαρίτσε. για την πολύ καλή διεξαγωγή της επίσκεψης. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μάθαμε. Και βεβαίω ε, υπήρξαν μια δυσκολίε σίγουρα λόγω των των συνθήκων τη επίσκεψή μα. Η επίσκεψη στα ορυχεία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και οι συζητήσεις πακολούθησαν. ακολούθησαν. Είχαμε άλλωστε προγραμματίσει να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η βιωσιμότητα, την εξαιρετική ε, βιομηχανία, τους ε, που ζουν στην περιοχή και θέλαμε να συλλέξουμε πραγματικά στοιχεία για αυτήν την επιχείρηση, την Latin American, την τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο εξόρυξης πλατίνας και είχα άλλωστε να είχα και κάποιες συναντήσεις, συναντήσεις από τα στοιχεία που συλλέξαμε βεβαιωθήκαμε για την ευθύνη και της BASF ε, σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης, χειρισμού των ε, ε ορικτών. Η δική μας ευθύνη για τους όρους παραγωγής, για τους τοπικούς πληθυσμούς, είναι να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα. Δεύτερο, για την ε, γεωργική μεταρρύθμιση. Η συζήτηση ήταν ε, πολύ έντονη. Η μεταρρύθμιση της χρήσης γης που κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει διότι διαφορετικά δεν θα καταστεί εφικτή η καταπολέμηση της φτώχειας που πλήττει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Αυτό συνδέεται και με το ξεπέρασμα των ε, καταλήπων του Απαρτχάιντ, ιδιαίτερο ρόλο εδώ παίζουν οι λευκοί γεωργοί, γιατί οι μαύροι γεωργοί δεν μπορούν ε, με τα μέσα που έχουν στα χέρια τους να ενισχύσουν την ε, ε, την παραγωγικότητα. Αυτό το επεσήμανε και η πρόεδρος του, της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Cape Town, η οποία και επισήμανε την ανάγκη ο πρόεδρος να εξασφαλίσει την ε, εφαρμογή της μεταρρύθμισης και νομίζω ότι και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει σαφές μήνυμα. Γεγονός είναι ότι δεν αρκεί να μιλάμε κάθε τρία-τέσσερα χρόνια για την ε, Νότια Αφρική. Αντιθέτως πρέπει και στο πλαίσιο του ε, διεθνούς εμπορίου να ε, καταστεί στρατηγικός μας εταίρος ο κύριο Κάμπελ Μπάνερμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές ε, αυτού του χρήσιμου ταξιδιού. Το πρώτο πράγμα που με εξέπληξε ήταν ε, η έκταση της ε, παραγωγής αυτοκινήτων στην ε, Νότιο Αφρική. Αυτοκίνητα τα οποία μάλιστα εξάγονται από, και προς το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ακόμη και προς τις ΗΠΑ. Είναι τεράστια αγορά εξαγωγέας. Το δεύτερο σημείο που με εξέπλησε, και αυτό είναι και παγκόσμιο δίδαγμα, είναι η κρατική παρέμβαση Ξαναλέω λοιπόν, ένα τέταρτο της συνολικής οικονομίας της Νοτιού Αφρικής έχει γίνει αντικείμενο ε, ιδιοποίησης από τον πρώην πρόεδρο, αυτό έχει πλήξει σημαντικότατα την οικονομία της χώρας, έχει δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα και για την ανάκαμψη της οικονομίας. Και τρίτον, μεταρρύθμιση της χρήσης γης. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα. Και εν ώψη του κινδύνου να γίνει μια δεύτερη Ζιμπάμπουε η χώρα, κάτι που θα ήταν καταστροφή για όλους, ο πρόεδρο ε, Ράμα Πόζα θεωρεί ότι με πολύ έξυπνο, θεωρώ ότι με πολύ έξυπνο τρόπο ε, χειρίζεται το θέμα, ε, πιέζει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της γης, του συστήματος χρήσης γης, δέχεται βεβαίως και μεγάλες πιέσεις, αν όμως παίξει σωστά τα χαρτιά του, θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να ωφελήσει τη χώρα και όχι να διώξει ε, ξένες επενδύσεις ο πληθυσμό τη χώρα έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα κατά 8% γιατί πολλέ ολόκληρε οικογένειε εγκαταλείπουν τη χώρα. Είναι κρίμα διότι η χώρα αυτή έχει πραγματικά τεράστιε δυνατότητε και είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ για τα στοιχεία αυτά που μας ε, μετέφεραν οι συμμετέχοντες στην αποστολή. Ευχαριστούμε την κυρία Σχάκε ως επικεφαλής θα παρακολουθούμε στενά το θέμα και στο μέλλον. Uh, Έχουμε ένα πρόβλημα διότι η Επιτροπή για το επόμενο σημείο δεν είναι εδώ. Θα περιμένουμε πέντε λεπτά. Okay. Three minutes break. Τρία λεπτά διάλειμμα. Okay, so, dear colleagues. Συνάδελφοι, σημείο 17. Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Στην τελευταία ομιλία του κυρίου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, εξεπλάγει για το γεγονός ότι ο κύριος Γιούνκερ ανακοίνωσε αυτή την νέα οπτική για την συγχώνευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης σε μια παναφρικανική συμφωνία σε ευθυγράμμιση με τις συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου με την Ήπειρο συνολικά. Αυτό δεν το περιμέναμε και ούτε είναι και ακριβώς σαφές τι εννοεί. Ιδίως για τα ΗΠΑ που μιλάμε, που συζητάμε εδώ και πώς μπορούν να ε, υλοποιηθούν όλα αυτά. Και υπάρχει αυτή η περιφερειακή προσέγγιση στις είπα διότι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό και από το ενδοαφρικανικό εμπόριο, γι' αυτό και την χάνει βεβαίως της υποστήριξής μας. Το σχέδιο όμως, με τον τρόπο που ανακοινώθηκε, ήταν κάτι νέο και έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο της Επιτροπής, η οποία και έχει το λόγο για 6 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη θέσπιση μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου που θα καλύπτει όλη την Αφρική μέσω της εμπορικής της πολιτικής, μεταξύ άλλων. Στην ομιλία της 12 η Σεπτεμβρίου, ο κύριος Γιούνκερ πρότεινε μια συμμαχία για τις βιώσιμες επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας και εδώ περιλαμβάνονται μια σειρά από σημαντικές ιδέες για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από το εμπόριο με την Αφρική. Μεταξύ των εργαλείων για την επίτευξη αυτής της επιτυχημένης ε, συμμαχίας είναι το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων και οι εμπορικοί κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο με την Αφρική. Κοιτάζοντας την ανακοίνωση, βλέπετε ότι τα εμπορικά καθεστώτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ως ε, δομικές μονάδες υπέρ της ε, ζώνης ελευθέρου εμπορίου της Αφρικανικής Υπήρου που βρίσκεται υπό οικοδόμηση. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επικέντρωση στην ε, εφαρμογή των ε, συμφωνιών οικονομικής ε, εταιρικής σχέσης στην υποσαχάρια Αφρική, την διεύρυνση των ΗΠΑ σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους τομείς της οικονομίας και την εντατικοποίηση των συνομιλιών με την Βόρεια Αφρική για τις ε, ολοκληρωμένες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή με την Τινησία στο, με το Μαρόκο στο μέλλον. Συνεχίζουμε επίσης την υποστήριξή μας άλλων δράσεων υπό την Συμμαχία, για τις οποίες δεν είμαστε αρμόδιοι εδώ στην, ε, εμείς στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, αλλά μπορώ να τις αναφέρω. Υπάρχει τεχνική και οικονομική συνδρομή στην ζώνη ελευθέρου εμπορίου της Αφρικανικής Υπήρου, την οποία διαχειρίζεται η DG DEFCO υπάρχουν σύμφωνα για την ανάπτυξη και την απασχόληση με την υποσαχάρια Αφρική στην εφαρμογή των οποίων θέλουμε να συμμετέχουμε και εμείς ως DG εμπορίου και που μας αφορούν ως θέματα γιατί αφορούν έγγραφα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους Αφρικανούς εταίρους μας να αξιοποιήσουν ε, τοπικές και παγκόσμιες αλυσίδας αξίας και να αξιοποιηθούν για τους τομείς προσθέμενης αξίας. Υπάρχει ένας διάλογος ε, με τους Αφρικανούς εταίρους μας, ο οποίος στόχο έχει να ενισχυθούν οι επενδύσεις, να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον και αυτό ε, εξυπηρετεί, αυτό το στόχο εξυπηρετεί και η task force που συνέστησε ο κύριος Χόγκαν. Η task force αυτή δημιουργεί κίνητρα που είναι αναγκαία για την προσέλκυση επενδύσεων στις αφρικανικές χώρες και περιφέρειες και γι' αυτόν τον λόγο ε, εντάσσεται υπό τον τρίτο πυλώνα του Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων που αυτή τη στιγμή συντάσσεται για τους Αφρικανούς εταίρους μας. Το εμπόριο επίσης πρέπει να συμπεριληφθεί ε, περισσότερο ε, στον δημόσιο διάλογο που έχουμε με μέσω του φόρουμ για, ε, για το αφρικανικό εμπόριο και τέλος τονίζουμε την υπόσχεση της συμμαχίας για ε, καλύτερη στόχευση της ανθρωπιστικής βοήθειας έναντι του εμπορίου, την βοήθεια ε, όσον αφορά κανονιστικά θέματα, προδιαγραφές ε, προϊόντων και βρισκόμαστε σε συνεχή και στενή συνεργασία με τους συναδέλφους μας από την DG ΔΕΦΚΟ για τα θέματα αυτά. Κυρία Ρέντα. Euh, Ευχαριστώ. Όπω και εσεί, Πρόεδρε, ξεπλάγει με τη δήλωση του κυρίου Γιούνκερ όταν ε, εκφώνησε την ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση και έχω διαφορετικά, διάφορα ερωτήματα να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την Αφρικανική Ήπειρο. Εάν ισχύει ότι η διπυρωτική αυτή περιοχή ελεύθερων συναλλαγών ε, υποστηρίζεται ανέκαθεν από την Ευρώπη, γιατί είναι σημαντικό να αναπτυχθούν και στην Αφρική οι συναλλαγές, οι ενδοαφρικανικές συναλλαγές, τότε θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ακριβώς στη δημιουργία αυτής της διπυρωτική ζώνης. Διότι πριν από μερικά χρόνια ήδη δεν μπορούσαμε να προωθήσουμε εσωτερικά τη δημιουργία εσωτερικών ε, ομάδων περιοχών στην Αφρική. Είχαμε αποτυχία των σχέσεων τερική οικονομική σχέση που αφορούσαν ομάδα χωρών. Η μόνη τέτοια σχέση και συμφωνία που μπόρεσε να ολοκληρωθεί ε, με κάποια περιφέρεια της Αφρικής ήταν η ΣΕΝΤΕΚ. Ως προς την Ανατολική Αφρική ή με τη Δυτική Αφρική το ίδιο και η οικονομική εταιρική σχέση με την Κεντρική Αφρική, που σήμερα δεν είναι καν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ε, έχουν παραμείνει κενό γράμμα, ε, κενό νοήματος κείμενο. Θα πρέπει λοιπόν τώρα ε, να δούμε τι μπορεί να γίνει με όλε τι αφρικανικέ χώρε. Αν και βέβαια μέχρι τώρα η σταδιακή μα έχει αποτύχει ω προ την περιφερειακή προσέγγιση. Πώ μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε τι θα συμβεί. Μου φαίνεται ιδιαίτερη κατάσταση και γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Trade τι μέσα έχουν πλέον στη διάθεσή τους για να μπορούν να προωθήσουν αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Αυτό που έθεσε επιτάπητος ο κύριος Γιούγκερ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι είδους ε, αντίθεση μπορεί να υπάρξει μεταξύ αυτής της προσπάθειας και της όλης διαπραγμάτευσης για την συμφωνία μετά την Κοτονού για να περιλαμβάνονται εκτός από την Αφρική και οι χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Άρα δεν είναι μόνο οι διαπραγματεύσει με τι αφρικανικέ χώρε που μα ενδιαφέρουν. Μήπω υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών στρατηγικών. Από τη μια, ένα ε, μια μεγάλη υπερμεγέθης εμπορική συμφωνία με την Αφρική και μετά το θέμα της Κοτονού. Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της συμφωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην συμφωνία ε, μετά την Κοτονού υπάρχουν πρώτα τρεις βασικές αξίες. Η ανάπτυξη, η διακυβέρνηση και το εμπόριο. Και τα τρία αυτά είναι άξονε που πάνε μαζί. Αυτό που έθεσε επιτάπητο ο κ. Γιούγκερ είναι λε και ενέκρινε στρατηγική τη Κίνα για εμπορικά θέματα. Εμπόριο σκέτο. Μόνο επιχειρήσει. Και ξέχασε λίγο του άλλου δύο θεμελιώδει πυλώνε τη διακυβέρνηση και τη ανάπτυξη. Διερωτώ με λοιπόν, η δήλωση Γιούγκερ που αγνοεί τους δύο αυτούς καθοριστικούς πυλώνες για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Τι θα γίνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θα με ενδιέφερε να μάθω από την Κομισιόν είναι το εξής. Στα κράτη-μέλη είδαμε και φέτος και πέρσι να θεσπίζονται και εθνικέ στρατηγικέ για την Αφρική ή τουλάχιστον να βρίσκονται στο στάδιο τη προετοιμασία. Ξέρω από τη Γερμανία ότι ε, χαράξαμε ένα σχέδιο Marshall για την Αφρική με ευθύνη του Υπουργού κ. Μούλερ αυτό που θα με ενδιέφερε είναι σε ποιο βαθμό οι εθνικές στρατηγικές, τα εθνικά σχέδια ε, βρίσκονται σε επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά ή πρόκειται απλώς για αυτό, αυτόνομη πορεία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που προτείνετε εσείς. Πρόκειται για αυτόνομη πορεία και στρατηγική για την Αφρική ή προσπαθείτε να εντάξετε σε αυτό και τις ήδη υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Ναι, ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία από τον κύριο Γιούνκερ και αναρωτιέμαι πόσο σε βάθος την είχε μελετήσει αυτή την πρότασή του ε, λαμβανομένου υπόψη ότι μιλάμε για πολύ διαφορετικές χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης από πολύ ε, χαμηλής ανάπτυξης χώρες μέχρι και μέσης ανάπτυξης. Πώς η Κομισιόν λοιπόν λαμβάνει υπόψη της αυτή την ποικιλομορφία ε, των χωρών της Αφρικής. Και είναι δύο ε, στοιχεία τα οποία λείπουν πολύ σημαντικά. Το πρώτο αφορά τη διακυβέρνηση. Οι παράνομες ε, ροές κεφαλαίου από την Αφρικανική Ήπειρο προς την Ευρώπη αλλά και προς άλλα μέρη του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι τριπλάσιες έως δι... δεκαπλάσιες από τις αντίστροφες ροές κεφαλαίου στην ε, Αφρικανική τι γίνεται λοιπόν με τη διακυβέρνηση. Ξέρω ότι υπάρχουν στην Αφρική μια σειρά από διαδικασίε που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των παράνομων κεφαλαιακών ροών. Νομίζω ότι ο Κόφι Ανάν ήταν πρόεδρος μιας σχετικής επιτροπής και ο πρόεδρος Μπέκι το ίδιο. Πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα στοιχεία για την ανάπτυξη Έχουμε πλέον το σχέδιο ε, εξωτερικών επενδύσεων. Πώς όλες αυτές οι διαστάσεις της βοήθειας και της ανάπτυξης θα εξασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση και άλλων τομέων όπως είναι η υγεία, η παιδεία που βοηθούν και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, για το εμπόριο. Υπάρχουν μηχανισμοί για να, βοηθηθεί, για να βοηθηθούν ε, περιφερειακές εμπορικές κοινότητες όπως στην ε, Δυτική Αφρική για παράδειγμα ε, έχετε κάποια διάσταση σε πιο περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την στρατηγική σε αυτά. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την ενημέρωση. Ο σκιώδης εισηγητής μας, η Λάουρα Σάντσες, δεν είναι εδώ. Ε, το συζητήσαμε όμως κάπως μεταξύ μας και εκτιμούμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ προσπάθησε να δημιουργήσει μια νέα μορφή σχέσεων με την ε, Αφρική το είπε στην παρουσίασή του. Αλλά όπως είπαν ε, και οι συνάδελφοι, πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά σε αυτήν τη συμφωνία σε θέματα εμπιστοσύνη. Δηλαδή να υπάρχει μια πιο συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Αυτό θα βοηθήσει. Και η Μαρία Ρένα ήδη ζήτησε τη διαδικασία μετά το Κοτονού με τους τρεις πυλώνες. Οπότε η ερώτηση είναι, φαίνεται πως η διακυβέρνηση, ο πυλώνας της διακυβέρνησης δηλαδή, αλλά και της ανάπτυξης, προβάλλονται λιγότερο για τις αφρικανικές χώρες ΑΚΕ. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο εμπόριο. Δεν πρέπει όμως να συνεχίσουμε business as usual, να καθίσουμε να προβληματιστούμε για το πώς προχωράμε. Και ρωτάω την Επιτροπή, αυτός ο προσανατολισμός των Αφρικανικών χωρών για να δημιουργήσουν κατά κάποιο τρόπο μια τελωνιακή ένωση μεταξύ τους, πιστεύετε ότι είναι κάτι εφικτό κάτω από τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν ε, σε αυτές τις χώρες. Και τι σημαίνει αυτό βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για μας. Πώς θα συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η λογική της Τελωνιακής Ένωσης είναι να μην μπορέσουν κάποιες αφρικανικές χώρες να αναπτύξουν τη δικιά τους οικονομία. Και έπειτα θα υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των Αφρικανικών χωρών. Δεν είναι όλες ίδιες και είναι δικιά μας ευθύνη να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και κατάλληλα να συνοδεύσουμε τη διαδικασία. Και κάτι ακόμα. Οι επενδύσεις στην Αφρική, και αυτό είναι το μάθημα που πήραμε σχετικά με την εξορρυκτική βιομηχανία. Οι επενδύσεις που δίνονται σε αυτές τις χώρες εξυπηρετούν πραγματικά την βιώσιμη ανάπτυξη εκεί. Από την πλευρά μας δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και δεσμευτικές προϋποθέσεις, υποχρεωτικές ρήτρε. τι κάνουμε εμείς, ε, η Βορειοαμερική κτλ. Οδηγεί πραγματικά σε αλλαγή τη σημερινής κατάστασης στις χώρες αυτές. Οι εθνικές στρατηγικές επίσης των αφορικανικών χωρών με το δικό μας SPG θα πρέπει να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι. Ευχαριστούμε. Κύριε Σκάβερν. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εννοείται ότι και εμείς χαιρόμαστε για την κατεύθυνση αυτή μείωση των φραγμών στο εμπόριο με την Αφρική και βοηθούμε έτσι με απασχόληση και επενδύσεις. Όμως, με ανησυχεί κάπως όλη αυτή η ιστορία για τις διαφορές μέσα στην Αφρική. Φυσικά είναι διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο. Η φτώχεια είναι μεγάλη όπου και αν πάτε. Πάντως, εγώ ε, συναντήθηκα με τον κύριο Φαντέμπη που είναι ο πρόεδρος ε, του Αφρικανικού Κοινοβουλίου και το θέμα της ε, ενιαίας τελωνιακής ένωσης το συζητήσαμε. Εγώ δεν θέλω μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική. Πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία. Υπάρχει η Νιγηρία, Μαρόκο ε, με ε, δικαστικές διαδικασίες που δεν υποδέχτηκε πολύ θετικά η Νότια Αφρική. Πάντως υπάρχει μια γενικότερη ατζέντα για να γίνει η Αφρική κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι έτσι μόνο περισσότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ναι, στο ελεύθερο εμπόριο και στις επενδύσεις παντού στην Αφρική, απασχόληση για να μειωθεί η μετανάστευση σε κάποιο βαθμό, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα εθνικά όρια και σύνορα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εγώ τώρα, λέει ο και πάλι, συγκεκριμένα, ποιο είναι το συγκεκριμένο καθεστώς αυτής της ε, Παναφρικανικής περιοχής ελεύθερου εμπορίου. Υπάρχει γενική συμφωνία, αλλά οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές. Τουλάχιστον δεν είναι ξεκάθαρες. Πότε περιμένετε εσείς να έχετε έναν τέτοιο χώρο ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική. Πότε θα πιστεύετε ότι θα γίνει πραγματικότητα και τι θα περιλαμβάνει. Πιστεύετε ότι μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στη Ρουάντα και την Νότια Αφρική, για παράδειγμα, είναι μια καλή ιδέα. πώς αυτό συνδέεται με τις συμφωνίες εταιρική σχέσης. Μήπως θα ξεχάσουμε τελικά τις συμφωνίες εταιρική σχέσης, δεν θα πραγματευόμαστε πια τέτοιες συμφωνίες, άπαξ και υπάρχει αυτός ο χώρος ελεύθερων συναλλαγών αφρικανικούς. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σας τις ερωτήσεις. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι πράγματι η δήλωση Juncker πρέπει να λεφτεί υπόψη σε κάτι μακροπρόθεσμο, μια προοπτική πολύ μακροπρόθεσμα. Προς το παρόν ε, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία σε επίπεδο υπήρου καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις προηγουμένως από αφρικανικής πλευράς καταρχήν. Ένας τέτοιος χώρος ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Σε κάποιες περιοχές της Αφρικής πράγματι τα πράγματα έχουν προχωρήσει περισσότερο από ό,τι αλλού. Το θέμα είναι οι ομόλογοι ε, από πλευράς Αφρικής θα αναγνωρίσουν ε, τη δυνατότητα η Αφρικανική Ένωση να αναλάβει διαπραγματεύσεις, να κάνει αυτή τη δουλειά. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Δεν το ξέρουμε. Όλες οι πλευρές πάντως δουλεύουν και μέρος της στρατηγικής είναι οι συμφωνίε εταιρική σχέσης, δεν είναι ασύμβατες, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή άνοιγμα στο εμπόριο. Οι συμφωνίε εταιρική σχέση έτσι κι φτιάχνουν μια περιφέρεια όταν πρόκειται για περιφερειακέ τέτοιε συμφωνίε. Μαρία Ρένα, πολύ σωστά είπατε ότι το Σαντέκ είναι η μόνη περιφέρεια εταιρική συμφωνία στην περιοχή Ε, Στη Νότια Αφρική συμμετέχουν τέσσερι χώρε Πρόκειται για υποπεριφερειακή συμφωνία σχέση και όχι περιφερειακή. Μπορεί να γίνει τέτοιο όμω στο μέλλον. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου συζητούμε την ευάθυνση της συμφωνίας αυτής και να συμπεριληφθούν και άλλα θέματα όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, οι επενδύσεις, μεταφορές κτλ. Όλα αυτά εξαρτώνται από τη βούληση και την επιθυμία των Αφρικανών εταίρων. Η ολοκλήρωση της Αφρικανικής Υπήρου δεν είναι μια διαδικασία της οποίας ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι αφρικανική υπόθεση. Οι αφρικανικοί παράγοντες έχουν απόλυτη κυριαρχία γι' αυτό. Εμείς απλώς στηρίζουμε την διαδικασία και με τα εμπορικά μας μέσα και μηχανισμούς, τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών κτλ προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση του ίδιου στόχου. Το θέμα είναι να έχουμε βάνθηση στις εμπορικέ σχέσεις υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, κάτι που αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την Αφρική. Δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούμε από την αναπτυξιακή συνεργασία ή από τη διακυβέρνηση. Όχι. Θα συνεχίσουμε να έχουμε την Αφρική ως προτεραιότητα και σε άλλες μας πολιτικές. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, για παράδειγμα. Υπάρχουν και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε θα έλεγα ότι, ναι, υπάρχουν πολλές προκλήσεις και μέσα στην Αφρική για τον χώρο ελεύθερων συναλλαγών. Το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα προσπαθούν να κυρώσουν κάποιες συμφωνίες πριν υπάρχει οποιοδήποτε διακανονισμό σε επίπεδο υπήρου ή και με εμάς. Πρώτα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πλήρως ο αφρικανικός αυτός χώρος ελεύθερων συναλλαγών. Μιλάμε δηλαδή για μια προοπτική πραγματικά πολύ μακροπρόθεσμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και η αξιολόγηση όσον αφορά το καθεστώς και την σχέση Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου και εταιρική σχέσης. Απάντηση από την Επιτροπή. Το συγκεκριμένο καθεστώς του χώρου ελεύθερων συναλλαγών της Αφρικής έχει ως εξής. 49 χώρες έχουν υπογράψει από τις 55. Κάποιες χώρες όπως είναι η Νιγηρία, η Τανζανία δεν έχουν υπογράψει ακόμα και προβληματίζονται για το κατά πόσο θα υπογράψουν ή όχι τη συμφωνία. Κάποιες χώρες έχουν ήδη κυρώσει τη συμφωνία και η φιλοδοξία τους ήταν μέχρι τα τέλη της χρονιάς 22 χώρες να έχουν κυρώσει. Άρα τότε θα αρχίσει να ισχύει ο χώρος ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική. Ακόμα όμως δεν είμαστε εκεί. Υπάρχουν ζητήματα που ακόμα πρέπει να περάσουν από την ε, διαπραγμάτευση πριν αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο Αφρικανικός χώρος ελεύθερων συναλλαγών. Πρόκειται για αποκλεισμό κάποιων προϊόντων, γιατί θέλουν το 90% του διαφρικανικού εμπορίου να ελευθερωθεί. Οπότε πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο 10%. Ακόμα δεν έχει γίνει διαπραγμάτευση από αυτού. Συνεπώς, θα έλεγα ότι ακόμα βρίσκεται σε ανάπτυξη το σχέδιο. Και οι επόμενες εβδομάδες, μήνες θα δείξουν πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά ξέχασα και κάτι άλλο και συγγνώμη γι' αυτό. Μια άλλη ερώτηση που κάνατε για τη διαδικασία μετά το κοτονού γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες, που συνδέονται όμως πράγματι. Αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με την ομάδα ΚΕ, που αποφάσισε το Μάιο να λειτουργήσουν ως διαπραγματευτική ομάδα μαζί. Στη δικιά μας τη δομή θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακοί πυλώνες για την Αφρική, Καρεβική και Ειρηνικό. Οπότε πρέπει να δούμε πώς βλέπουν και αυτοί το θέμα. Η εντολή ΑΚΕ, αυτή καθεαυτή, αναφέρει ενδεχομένω περιφερειακούς πυλώνες στο μέλλον. Οπότε στόχος μας είναι να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε επ' αυτών το 2019. Άρα το πρώτο βήμα είναι οι χώρες ΑΚΕ υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί θα συνδεθούν οι περιφερειακοί πυλώνες. Οι περιφερειακοί πυλώνες πάντως είναι στα χέρια των περιφερειών ακριβώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτεί με τις περιφερειακές ομάδες χωρών. Εφόσον βέβαια είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τέτοια διαπραγμάτευση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πολύ μακροπρόθεσμη προοπτική. Πολύ ευχάριστο αυτό. Επόμενο σημείο, 18 και 19 μαζί. εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή τη δασική νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο. Ο λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ για την λεύκανση ξυλίας, το ξέπλυμα ξυλίας. Έχουμε ακούσει για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλά όχι για, για το ξέπλυμα ξυλίας που προέρχεται από την Ανατολική Ασία, δηλαδή την νομιμοποίηση των ε, προσόδων από την ξυλία. Υπάρχουν φοβερές ροές και συναλλαγές τέτοιου είδους στην Ανατολική Ασία με πρώτες ύλες από το Καμερούν, την Καμπότζη, το Λάος μέχρι που το Λάος απαγόρευσε τις εξαγωγές ε, πωλήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και την Κίνα, κατά κύριο λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ υπέγραψαν στις 19 Οκτωβρίου μια εθελοντική συμφωνία ώστε να περιοριστούν οι εξαγωγές προς άλλες χώρες. Η υπογραφή είναι το πρώτο βήμα μιας ε, μακράς διαδικασίας και είναι βεβαία ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα παρακολουθούμε διαρκώς το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία από την ε, υπογραφή και την κύρωση της εταιρική συμφωνίας με το Βιετνάμ μέχρι την υλοποίηση. Μέχρι το πρόγραμμα να είναι τόσο επιτυχές που το Βιετνάμ θα μπορέσει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις λεγόμενες άδειες FLECT Τι επικυρωμένε άδειε αυτέ με τη σφραγίδα τη νομιμότητα τέλο πάντων, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ως προς την όλη προσπάθεια πρέπει να προβλέψουμε μια πολιτική ώστε να μην εξάγεται παράνομη ξυλία προς τέτοιες χώρες, ιδίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα διασύνδεση με την Συμφωνία Ελεύθερου μπορείου που και αυτή συζητιέται εδώ. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Σαχραντήλ, τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, διότι είναι αξιοσημείωτο το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης στην ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου κάνει άμεση μνήμα στην ε, Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Είναι τόσο σύντομη φράση θέλω να τη διαβάσω. Κάθε μέρος θα ενθαρρύνει την πρόθεση και την εμπορία ανθρώπων, ε, προϊόντων συγγνώμη, από δάση που προέρχονται από τη βιώσιμη και νόμιμη δασοκομεία και ξυλία. Και αυτό θα αφορά το εμπόριο, τη διακυβέρνηση και την δασοκομεία ε, με τις λεγόμενες άδειε FLECT. Να τονίσω ότι με αυτή την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση που θα κρατήσει κάποια χρόνια, ελπίζουμε, και θα οδηγήσει στις άδειε FLECT των προϊόντων της δασοκομείας και ξυλία από το Βιετνάμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και ζητά καλύτερη διακυβέρνηση σε πολλούς τομείς στη χώρα στο Βιετνάμ συγκεκριμένα. Ουδέποτε δεν είδαμε να υπάρχει τόσο πολύ συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στο Βιετνάμ όσο στα πρώτα στάδια της υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν πολλές απαιτήσει για την αντιμετώπιση της διαφορά, διαφθοράς, η οποία ιδίω στα τελωνιακά είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και είναι καθοριστική σημασία για τις ροές ξυλίας από την Καμπότζη προς το Βιετνάμ κατά κύριο λόγο. Και νομίζω ότι τώρα που αποφασίσαμε να εγκρίνουμε τη σύσταση για την εθελοντική συμφωνία, καλό θα ήταν να <clears throat> συνοδευτεί και από ένα ψήφισμα αυτό. η ιδέα μου, και σας το προτείνω συνάδελφοι, είναι να θέσουμε κάποιους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης για να τους ε, αξιοποιήσουμε μέχρι τη φάση της κύρωσης που είναι κέρια για το Ευρωκοινοβούλιο και πριν την υλοποίηση της ε, εθελοντικής συμφωνίας. Διότι η πρόβλεψη των αδειών φλεκτ που είναι ο τελικός στόχος, θα γίνει με κατεξοδότηση πράξη. Άρα σας καλώ να κοιτάξετε το πολύ ενδιαφέρον αυτό εργαλείο το οποίο έχει δώσει ήδη κάποια αποτελέσματα με την Ινδονησία. Είναι η πρώτη χώρα που έχει άδειε φλεκτ, αλλά υπάρχουν κι άλλε. και σε όλε τι χώρε. Οι άδειε φλεκτ έχουν πολύ καλά, καλές επιπτώσεις στη διακυβέρνηση, τη βιωσιμότητα και το εμπόριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Αφού είστε και από τη Φινλανδία, είστε πλέον αρμόδια να μιλάτε για δάση, τη δασοκομεία. Έχετε γίνει διάσημοι παγκοσμίω. Ξέρετε ποιος είναι διάσημος για, την, για τον καθαρισμό των δασών. Η κυρία Ρενά, ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Συνολικά πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με τα διάφορα επιχειρήματα που υποστηρίχθηκαν. Υποστηρίζουμε τις συμφωνίες εθελοντικής εταιρικής σχέσης όπως με το Βιετνάμ για να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη ξυλία και αυτή η εταιρική σχέση FLEG θα βελτιώσει και την διακυβέρνηση, την δασοκομεία συγκεκριμένα. Με μια ιδιαίτερη μερίμνα για την κοινωνική διάσταση, της προκλήσει που αντιμετωπίζουν ε, οι μικρές βιτεχνίες επεξεργασία του προϊόντων ξυλία διότι δεν θα πετύχουμε την αποτελεσματικότητα που θέλουμε τις ρυθμίσεις μας αν δεν το κοιτάξουμε και αυτό. Το Βιετνάμ εισάγει ήδη κομμένη ξυλία, τεμάχια ξύλου από γειτονικέ χώρες όπως η Καμπότζη και το Λάος. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικές αρχές να γνωρίζουν την περιφερειακή διάσταση του προβλήματος και να λάβουν και τα απαραίτητα μέτρα. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε κάτι ανάλογο όπω την εθελοντική εταιρική σχέση με το Βιετνάμ και στι υπόλοιπε συμφωνίε μα που έχουμε υπογράψει και ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο λόγου χάρη. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ απελευθερώνει πλήρω το εμπόριο ε, προϊόντων ξυλία από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ. Το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συμφωνία αυτή, που προσεγγίζει την εμπορία των παράνομων προϊόντων ξυλία, δεν είναι αρκετά φιλόδοξο ακόμα δεν είναι δεσμευτικό. Οπότε, καλό θα ήταν να είμαστε συνεκτικοί σε σχέση με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτή η εθελοντική διαδικασία που επιτρέπει να επιτελεστεί κάποια πρόοδο, όμω πρέπει να έχουμε κατανάλογα εργαλεία. Να ε, υποχρεωθεί το Βιετνάμ να σεβαστεί τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει στα πλαίσια τη εμπορική του συμφωνία. Το ίδιο και για την περιφερειακή διάσταση. Υπάρχει και εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και το υπογράμμισε και η συγγετρία και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δηλαδή, η εφαρμογή η απαγόρευση μάλλον στο Βιετνάμ των παράνομων ε, εισαγωγών ξυλία, κυρίω από την Καμπότζη. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία και επιπλέον ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τι ροέ παράνομη ξυλία και προϊόντα παράνομη ξυλία στην Νοτιοανατολική Ασία, η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν εδώ ρόλο να παίξουν. Είναι η βασική υπεύθυνη για την νομιμοποίηση παράνομη ξυλία και των Στην Ιαπωνία είδαμε ότι υπάρχει προσπάθεια βελτίωση τη Ιαπωνική νομοθεσία ω προ τη διαχείριση τη παράνομη ξυλία στην χώρα. Όμω, ο νόμο που ψηφίστηκε είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα. Η μελέτη αντικτύπου που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι 25% των φορέων που έχουν σχέση με την εφαρμογή του νόμου δεν ε, ελέγχουν την νομιμότητα των προϊόντων ξυλία που φτάνουν στην Ιαπωνία. Άρα και η εμπορική συμφωνία που έχουμε με την Ιαπωνία θα πρέπει να μα κάνει να είμαστε σε επιφυλακή ε, σε σχέση με την εισαγωγή παράνομων προϊόντων ξυλία στη χώρα αυτή, ε, εφόσον ξέρουμε ευθύ εξ αρχή ότι η συγκλασιμότητα δεν εξασφαλίζεται στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή. κυρία Λαλόντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ την Χαϊντή Ναουτάλα για το εγγραφό τη. και συμφωνώ με τις συστάσεις της. Η ρύθμιση Fletched δείχνει ότι μπορούμε να συμφιλιώσουμε το εμπόριο με την προστασία του περιβάλλοντος και ελπίζω να υπάρξουν τέτοιες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλους κλάδους. Ε, η δασοκομεία είναι πολύ σημαντική για το Βιετνάμ. 45% της επικράτειας καλύπτεται από καλλιέργειες ή από δάση και είναι πολύ σημαντική για την τοπική οικονομία. Συνεπώς, πρέπει η εκμετάλλευση των δασών και της ξυλίας να είναι κάτι το βιώσιμο. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα καλό κείμενο και εννοείται ότι θα συστήσω στην ομάδα μου να το υπερψηφίσει. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Χέντι που μιλάει για την εφαρμογή, δηλαδή πώς θα είναι και ρεαλιστική και αποτελεσματική. Γι' αυτό έχω να συμπληρώσω με κάποιες ιδέες, ας πούμε για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις χώρες που έχουν μια συμφωνία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πώς ε, θα προχωρήσουν. Να ξέρουμε ότι η Κίνα που συνορεύει με το Βιετνάμ επηρέαστε πολύ από αυτό το φαινόμενο της παράνομης ξυλίας και θα ήταν μεγάλη νίκη αν μπορούσαμε να τη συμπεριλάβουμε και αν μπορούσαμε να έχουμε μια παγκόσμια ρύθμιση από αυτού. Έπειτα η υπεργολαβία πρέπει να μας απασχολήσει για τρίτες χώρες ώστε να μην υπάρχουν κενά τελικά στην ρύθμιση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Η Ανμαρή Μινέρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Χωτάλα για το άγραφο εργασία τη για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Αν θέλουμε εμπόριο με το Βιετνάμ, είναι πολύ σημαντικό το σύστημα αυτό εντοπισμού της παράνομης ξυλίας να λειτουργεί και να πιέσουμε το Βιετνάμ να τηρεί τις υποχρεώσεις του, τις δέουσας επιμέλειας δηλαδή. Η νομοθεσία του Βιετνάμ δεν φτάνει για την καταπολέμηση της παράνομης ξυλίας και υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει η ξυλία αυτή και στις ευρωπαϊκές αγορές. Με την παράνομη ξυλία δηλαδή από την Καμπότζη που μέσω Βιετνάμ μπορεί να φτάσει σε εμά. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Και να πιέσουμε επίσης και για μια πιο ευρύτερη οργάνωση προκειμένου να υπάρξει εφαρμογή της συμφωνίας από το Βιετνάμ αλλά και παγκοσμίω. Γιατί αυτό βοηθάει φυσικά την κοινωνία των πολιτών. Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με το Βιετνάμ αλλά και με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε εμά πρέπει να ενισχυθεί. Πιέζω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα και να ενημερωνόμαστε. Ευχαριστώ ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Άστριτ Σούμαρκερ είναι μαζί μας, Διευθύντρια για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ και που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμφωνούμε με όλα. Θέλουμε να τονίσουμε και εμείς αυτό που τόνισε η κυρία Χάουταλα, ότι το Βιετνάμ βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο ε, της παγκόσμιας ε, παραγωγής ξυλίας. Ήταν εκθετική η ανάπτυξη ε, των εισαγωγών και των εξαγωγών ξυλίας στην χώρα αυτή και εισάγει και εξάγει λοιπόν στις μεγαλύτερες αγορές η Βιετνάμ. Αυτό βεβαίως δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία, τους σωστής ε, κανόνες, ακριβώς γιατί είναι κομβική σημασία στο Βιετνάμ για την καταπολέμηση του λαθρεμπολίου λαθρεμπορίου ξυλίας. Η κυρία Χάουτελα περιέγραψε ε, λεπτομερώς και πολύ καλά τους στόχους. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θέλω απλά να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, σημασία της περιφερειακής διάστασης. Αυτό ε, δεν μπορεί κανείς παρά να το τονίζει. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με το Βιετνάμ. ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Λάος, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Μιανμάρ. Σε διάφορα επίπεδα βεβαίως και με διαφορετική πρόοδο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί το Βιετνάμ ώστε να ενισχυθούν οι διατάξεις νομιμότητας ε, ε, στις χώρες από τις οποίες εισάγει ξυλία ε, το Βιετνάμ. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα η πολύ ανησυχητική κατάσταση γύρω από την Καμπότζη. Εμείς συζητούμε το θέμα αυτό με τις βιετναμέζικες αρχές, γνωρίζουν βεβαίως το θέμα, γνωρίζουν και το έργο της, ε, του Οργανισμού Περιβαλλοντικών Ερευνών που ε, θέτουν αυτούς σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση του έργου τους Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανησυχητική, η προβληματική κατάσταση με την ε, Καμπότζη. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, τα οποία όμως ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Η κύρωση είναι, από πλευρά Βιετνάμ ε, της συμφωνίας είναι μια πρώτη κίνηση που ε, δείχνει την προθυμία του Βιετνάμ να δημιουργήσει ένα πραγματικά νόμιμο, ασφαλές σύστημα. Στην πορεία των χρόνων θα φανεί αν πράγματι θα αποκομίσουμε τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε και ε, βεβαίως όπως είπε η κυρία Μινόρ είναι πολύ σημαντικό το σύστημα της δέωσας επιμέλειας και χαιρετίζουμε την ε, πρόταση της Κομισιόν ότι η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά μια αντιγραφή επικόλυση άλλων συστημάτων ή διαδικασιών, αλλά να είναι μια πραγματικά ουσιώδης διαδικασία η οποία θα εξασφαλίζει ότι θα καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο ε, και αποτελεσματικό σύστημα. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Το Βιετνάμ έχει λάβει ήδη μέτρα προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία και η παραγωγή ξυλίας αλλά και η οργανώση κοινωνίας των πολιτών και σε συνεργασία με το Βιετνάμ θα ε, προχωρήσουμε και βεβαίως σε αξιολόγηση του συστήματος και όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αυτή βεβαίω θα υποβάλουμε και πρόταση κατεξοδότηση κανονισμού. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην εργασία και με τους μεγαλύτερους εισαγωγείς, είπα, Κίνα, με την Κίνα υπάρχει και ένας διμερής μηχανισμός συνεργασίας και ε, εμείς ανησυχούμε και του το έχουμε δηλώσει για την ε, πιθανή εισαγωγή παράνομων προϊόντων ξυλίας στην Κίνα και από εκεί ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε και έχουμε παρακινήσει τους Κινέζους ομολόγους μας να θεσπίσουν πιο δεσμευτική νομοθεσία. Βεβαίως είναι σχετικά πρόσφατη η νομοθεσία τους, οπότε είναι δύσκολο να ξαναμπούν σε μια διαδικασία άμεσης τροποποίησης, αλλά τουλάχιστον στο, ε, ε, στο, στην Ιαπωνία ε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα προαιρετικά, τα εθελοντικά μέτρα γενικά γίνονται πιο σεβαστά, τηρούνται περισσότερο από ό,τι σε, ε, σε άλλα μέρη του κόσμου, σε άλλες χώρες του κόσμου. Αυτά από πλευρά μα. Σα καλώ όλου να υποστηρίξετε τη συμφωνία αυτή, γιατί πραγματικά ε, θα είναι εξαιρετικό εργαλείο στην προσπάθειά μα να καταπολεμήσουμε την, ε, το λαθρεμπόριο ξυλία. Ευχαριστώ πολύ, Χάιντι. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που έκαναν οι σκιώδεις συζητητές. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν για το έργο της, για αυτό το πολύ σημαντικό μέσο. Γιατί χρειάστηκε σημαντική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, εμπορίου, περιβάλλοντος ε, και άλλων και νομίζω ότι και εμείς από πλευράς ε, Κοινοβουλίου μπορούμε να ενισχύσουμε το έργο αυτό. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικό έργο. Είναι ε, πολύ θετικό το γεγονός ότι... Ε, προτάθηκε μέσω τροπολογίας να αναφερθούν και ορισμένε βέλτιστες πρακτικές. Αν Μαρή, έκανες μια πολύ σημαντική παρατήρηση για το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής για την αποτροπή εισαγωγής λαθρέων προϊόντων ξυλίας. Προϊόντων που προέρχονται μάλλον από ε, λαθρεμπόριο ξυλίας. Είναι σημαντικό λοιπόν το Βιετνάμ να θεσπίσει νομικά μέτρα που θα αποτρέπουν πλήρως την εισαγωγή ε, λαθρέων παράνομων προϊόντων ξυλίας στην επικράτειά του προκειμένου να μην επανεξάγονται στη συνέχεια σε άλλες αγορές. Θα γίνει και μια διερευνητική επίσκεψη τον Ιανουάριο είναι σημαντικό για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα επί τόπου. Μετά την διακοπή για τα Χριστούγεννα θα σας δώσω περισσότερες πρακτικές λεπτομέρειες για το ποια στοιχεία θα εντάξουμε τελικά στο ψήφισμα, αλλά θέλω από σήμερα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε να καταλήξουμε σε ψήφισμα, γιατί είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο προκειμένου να προσθεθούν στη συμφωνία κάποιοι συγκριτικοί δείκτες. Γνωρίζω ότι κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις θεωρούν ότι το VPA δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο γιατί το Βιετνάμ δεν είναι έτοιμο, αλλά όπως είπε και η Κομισιόν θεωρώ και εγώ ότι βρισκόμαστε απλά στην αρχή μιας διαδικασίας που θα είναι μακρά και που ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει τόσο τη χώρα του Βιετνάμ όσο και τα παγκόσμια δάση. Ευχαριστώ. Μεγάλος ο δρόμος μπροστά μας. Είμαστε στην αρχή, λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε εδώ στο θέμα αυτό στην Επιτροπή τον Ιανουάριο και καλή επιτυχία στο ταξίδι σας στο ε, Βιετνάμ. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα σημεία 18-19. Το, 20, το σημείο 20 θα το συζητήσουμε μαζί με την Επιτροπή ΔΕΒΕ στην αίθουσα PH4 Β 1. Μεταφερόμαστε στην αίθουσα εκείνη για τη συνέχιση της συνεδρίασης της Επιτροπής μας.